Uh, chers collègues, ladies and gentlemen, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Το πρώτο σημείο μας είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη? Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 5ης και 6ης Νοεμβρίου 2014. Θέλετε να προσθέσουμε, να αλλάξουμε κάτι στα πρακτικά αυτά μήπως? Όχι, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχουμε δηλαδή τίποτα για το σημείο 3. Σημείο 4. Θα δώσω το λόγο στην Μανουέλα Σάμεκ. Πρόκειται για την αξιολόγηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 στο πλαίσιο της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και ολίγοι κύριοι, καλό απόγευμα. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της μελέτης αυτής που κάναμε εμεί όσον αφορά τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε τη μελέτη αυτή για να βοηθήσουμε την Επιτροπή σας να αξιολογήσει την στρατηγική προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της πλατφόρμας του Πεκίνου. Η αρχική ιδέα ήταν επίσης να γίνει η αξιολόγηση αυτή ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις όσον αφορά την μελλοντική στρατηγική για μετά το 2015. Εδώ έχετε βέβαια την σύνθεση, αλλά νομίζω ότι έχετε και την μελέτη, μάλλον θα την έχετε σε λίγες μέρες. Ε, χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η αξιολόγηση της πολιετούς πολιτικής, του πλαισίου πολιετούς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την στρατηγική στα πλαίσια αυτού του πλαισίου πολιτικής. Επικεντρωνόμαστε στη σχέση κυρίως της στρατηγικής 2010-2015 με τους στόχους της πλατφόρμας του Πεκίνου και τις άλλες δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στον τομέα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την αξιολόγηση της στρατηγικής. Λαμβάνει υπόψη τα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα η στρατηγική σε σχέση με τους στόχους της πλατφόρμας του Πεκίνου και εξετάζει και όλα και όλες τις άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην εσωτερική και εξωτερική συνοχή της πλατφόρμας ή μάλλον διορθώνω μελήτρια της στρατηγικής. Κατά πόσο δηλαδή η στρατηγική καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εξετάζει κατά πόσο υπάρχει συνοχή μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Επίσης εξετάζει και την εξωτερική συνοχή, συνοχή δηλαδή με άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των δύο φύλων και εξετάζει και την εφαρμογή της στρατηγικής. Τι έγινε δηλαδή και αν υπάρχουν επιπτώσεις και αξιολόγηση, σύστημα αναφοράς όσον αφορά τα αποτελέσματα της στρατηγικής. Το τρίτο κεφάλαιο τα βάζει όλα αυτά μαζί και καταλήγει σε κάποιες συστάσεις για βελτίωση όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική. Λέει τι θα μπορούσε να γίνει για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ακόμα αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής. Η αξιολόγηση πρέπει να ξέρετε ότι βασίζεται ιδιαίτερα σε αξιολογήσεις, σε έρευνες, σε μελέτες Έχουμε επίση προχωρήσει και σε κάποιες συνεντεύξεις. Δυστυχώς δεν είχαμε πολύ χρόνο για την μελέτη αυτή, οπότε είναι λίγες οι συνεντεύξεις. Και τελικά υιοθετήσαμε μία πολιτική ανάλυση και αξιολόγηση για να καθορίσουμε την μελλοντική μας προσέγγιση. Θα συνοψίσω τώρα τα κύρια στοιχεία και τις αδυναμίες που εντοπίσαμε αναλύοντας τα έγγραφα αυτά και αναλύοντας ε, την στρατηγική 2010-2015. Επίσης θα αναφερθώ και στις συστάσεις που πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μελλοντικής στρατηγικής. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία. Πρώτον, το πρώτο σημαντικό είναι η έγκριση μιας διτής προσέγγισης που βασίζεται και σε ειδική δράση για την ισότητα των φύλων, αλλά και για την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα θέματα που εξετάζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και χώρες μέλη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πιστεύουμε ότι είναι ο εντοπισμός προτεραιοτήτων, που δηλαδή πρέπει να επικεντρωθεί η στρατηγική οι πέντε κύριες προτεραιότητες δηλαδή στις οποίες βασίζεται η στρατηγική. Όσον αφορά την καταλληλότητα της στρατηγικής σε σχέση με τις ανάγκες που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, εμείς πιστεύουμε ότι οι προτεραιότητες και οι δράσεις που αναφέρθηκαν ήδη το 2010 στη στρατηγική είναι κατάλληλες, είναι οι σωστές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνεπώς έγινε μια επιλογή ώστε να επιλεχθούν οι πιο κατάλληλες τα πιο κατάλληλα στοιχεία και οι πιο κατάλληλες προσεγγίσεις. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του στρατηγικούς στόχους της πλατφόρμας του Πεκίνου. ιδίω για θέματα που είναι πολύ σημαντικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή γυναίκες και οικονομική εξουσία, εκπαίδευση και κατάρτιση, καταπολέμηση της οικογενειακής ε, βίας, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, θεσμικοί μηχανισμοί, προκειμένου να προωθηθεί η άνοδος των γυναικών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Αναφέρονται και άλλα σημεία που συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του Πεκίνου. Αλλά αυτά είναι που σας είπαν τα πιο σημαντικά, τα άλλα ίσως έχουν λιγότερη σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η στρατηγική πέτυχε πολλά, πολλούς από τους αρχικούς στόχους που ήθελε να πετύχει. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνδυτοποίηση, δράσεις δηλαδή συνδυτοποίησης του κόσμου, όσον αφορά τη δημιουργία ιστοσελίδων, οδηγιών, κατευθυντηρίων γραμμών, μελετών, ερευνών. Ε, φτιάχτηκαν εργαλειοθήκες, υλικό για κατάρτιση και ιδιαίτερα, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είχαμε και την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την συλλογή δεδομένων. Το έρος που να ξέρετε ότι τώρα ε, περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία αναφύλλω και μας δίνει πληροφορίες για πολύ σημαντικά ζητήματα. Σε σχέση με την ισότητα βέβαια πάντα. Και μάλιστα όχι μόνο η Eurostat αλλά και άλλοι οργανισμοί και το FNA και άλλοι κάνουν έρευνες, μελέτες, κάτι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι γίνεται όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πράγματα τα οποία πριν από μερικά χρόνια δεν λαμβάνονταν καν υπόψη. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Είναι χάρη στη στρατηγική που το πετύχαμε. Έχουμε και νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα τα οποία προωθήθηκαν στα πλαίσια της στρατηγικής, ακόμα και αν μερικές φορές ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε νομοθεσία για πολλά ζητήματα. Τώρα, ποιες είναι οι δυναμίες και τα εμπόδια. Η δράση που αναφέρεται στη στρατηγική εντοπίζει γενικά, όχι όμως συγκεκριμένους στόχους με χρονοδιάγραμμα για το πότε θέλουμε να πετύχουμε τον κάθε στόχο ή ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της μίας ή της άλλης δράσης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σαφή ένδειξη και ανάθεση ευθυνών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Υπάρχουν βέβαια κάποιες νέες προκλήσεις που αναπτύχθηκαν όσο προχωρούσε η στρατηγική. Νέες προκλήσεις σημαντικές και που πρέπει να τις συμπεριλάβουμε και στη μελλοντική στρατηγική. Για παράδειγμα, όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού. οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι φιλικού γένους, είναι γυναίκες που ζουν με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχει, υπάρχουν ε, προβλήματα που έχουν να κάνουν ε, με τις μεταναστευτικές ροές. Και εδώ υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Να λοιπόν πράγματα τα οποία θα έπρεπε επίσης να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική. Και υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα των συνεπειών της μακροχρόνιας πια οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στους άντρες και στις γυναίκες. Ενώ για τους άντρες οι επιπτώσεις φάνηκαν αμέσως, αμέσως η κρίση είχε επιπτώσεις απάνω τους, γιατί έχασαν τη δουλειά τους πολλοί άντρες. Για τις γυναίκες όμως τα αρνητικά της κρίσης αυτής τώρα αρχίζουν να φαίνονται. Και θα φανούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Γιατί οι γυναίκες θα επηρεαστούν περισσότερο από τις περικοπές στους προπολογισμούς, από τα δημοσιονομικά μέτρα κλπ. Γιατί συνήθως το πρώτο το οποίο κόβεται είναι τα κοινωνικά επιδόματα. Άρα λοιπόν και πάλι οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες θα επομισθούν το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας για την οικογένεια με λιγότερα χρήματα. Επιτόλες οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα των συντάξεων, οι αλλαγές στο κράτος ευημερίας ή στην κοινωνική προστασία, είχαν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στους άντρες και στις γυναίκες. Και είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό πριν εφαρμόσουμε τέτοιες πολιτικές. Δηλαδή από πριν να ψάξουμε να δούμε τι διαφορές θα υπάρχουν στις επιπτώσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε και ποιος είναι αυτός ο οποίος τελικά θα πληρώσει περισσότερο για τέτοιες πολιτικές. Ένα άλλο πρόβλημα, μια άλλη αδυναμία είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και αξιολόγηση της πρόοδου της στρατηγικής. Υπάρχει μια ομάδα η οποία αποτελείται από ανθρώπους από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που ελέγχουν τι κάνουν οι γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά δεν είναι ένα σύστημα αυτό καθεαυτό που να συγκεντρώνει δεδομένα, που να έχει δείκτες και άρα δεν γίνεται τελικά αξιολόγηση συνολική μέχρι τώρα για το τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και τι επιπτώσεις είχε. Η Υπάρχουν επίσης και περιορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά ε, την διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Ιδιαίτερα σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Περιβάλλον, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες διεθνές εμπόριο, μακροοικονομικές πολιτικές, δημοσιονομικές πολιτικές, μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν πολλές βιομηχανικές πολιτικές, τέλος πάντων πάρα πολλοί τομείς πολιτικής όπου δεν υπάρχει ενημέρωση και συνδυτοποίηση για το ότι χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας τη διάσταση του φύλου. Η οποία τι μας λέει, μας λέει ότι η κάθε πολιτική μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στους άντρες και διαφορετικές στις γυναίκες. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το ξέρουμε και να το αξιολογούμε, να το μετράμε για να καθορίσουμε τις επιλογές μας στους τομείς αυτούς πολιτικής. Από την άλλη μεριά γίνονται πολλά για την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οπότε, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το gender mainstreaming, τη διάσταση αυτή του φύλου δηλαδή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές. Και το άλλο βέβαια είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020, που δεν αναφέρεται ρητά η στρατηγική. Άρητα ναι, αναφέρονται οι πέντε εμβληματικές δράσεις που μιλάνε και για την ισότητα, αλλά δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορα εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν την εφαρμογή της στρατηγικής. Το ένα είναι η έλλειψη των πόρων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και οικονομική, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική. Υπάρχει η μονάδα ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχει αρκετούς πόρους. Είναι αδύνατον με τόσο λίγους ανθρώπους, όσο αφοσιωμένοι και να είναι, δεν είναι δυνατόν να μπορούν και να πιέσουν για την καλή εφαρμογή της στρατηγικής αυτής σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Και μιλάμε τώρα για μία μονάδα μέσα σε όλες αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Που πώς να έχει τη δύναμη να πιέσει τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις να λάβουν και εκείνες υπόψη τους τη διάσταση του φύλου στη λήψη αποφάσεων στους δικούς τους τομείς. Και το άλλο πρόβλημα είναι η μειωμένη θεσμική δυνατότητα. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι είναι δύσκολο για μία μονάδα μιας μόνο γενικής διεύθυνσης να μπορεί να πιέσει όλες τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις να κάνουν το ίδιο. Να λάβουν υπόψη τους τη διάσταση του φίλου, Δεν έχουν αρκετή δύναμη γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την σύντομη περίληψη που σας έκανα για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της στρατηγικής, τι ενδείξεις έχουμε τώρα συμπεριλάβει στην έκθεσή μας τις συστάσεις. Κάποιες ε, μιλάνε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη σημασία που έχει η στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, έτσι, γιατί υπάρχει η στρατηγική του 2020 και άρα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της στρατηγικής αυτής στα πλαίσια όλων των άλλων των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα στοιχείο λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς πολιτικής που είναι σημαντικοί για την ισότητα των δύο φύλων και στα πλαίσια της απασχόλησης και ε, της ε, συμμετοχής στην κοινωνία. Πριν σας μίλησα για τις συντάξεις, για τα ασφαλιστικά κλπ. και στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων αλλά και εκτός απασχόλησης και κοινωνικής διάστασης. Είπαμε, είναι το περιβάλλον, οι οικονομικές πολιτικές, η επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ε, μεταφέρουν στερεότυπα. Ακόμα και για τις μεταφορές πρέπει να λαμβάνετε υπόψη διάσταση του φύλου. Στον προπολογισμό, γιατί εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Πέρυσι κάναμε μία μελέτη για την Επιτροπή ΦΑΜ για να δούμε η διάσταση αυτή του φίλου πόσο λαμβάνεται υπόψη στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για παράδειγμα. Κανένας δεν σκεφτόταν το θέμα της διάστασης του φύλου όταν παίρνανε αποφάσεις για τον προϋπολογισμό. Και όμως υπάρχουν μέσα για αυτή τη δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι ένα Παράδειγμα, το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη στοιχείων, δεδομένων και έρευνας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Συχνά βλέπετε, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι σαφές πώς θα εξετάσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων σε άλλους τομεί πολιτικής. Στις μεταφορές για παράδειγμα, πώ το κάνεις αυτό, στο περιβάλλον ή στη βιομηχανική πολιτική. Και όμως είναι δυνατόν να δούμε πώς διαφορετικές επιλογές σε αυτούς τους τομείς μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άντρες. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερη έρευνα, περισσότερα δεδομένα και δείκτες. Άρα πρέπει να επενδύσουμε για να τα έχουμε αυτά. είναι κάτι που έχει αρχίσει. Και είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής και αυτό, αλλά θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να αρχίσουμε να απευθυνόμαστε στους άντρες. Περισσότερο από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και στους άντρες και στις γυναίκες βέβαια. Για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία σε βάρος των γυναικών. Ποια είναι η ανάμειξη των ανδρών στην πρόληψη, στη συνειδητοποίηση. Είναι πολύ σημαντικός. Αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών είναι περισσότερο πρόβλημα των ανδρών παρά των γυναικών. Συνεπώς οι άντρες πρέπει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Άρα πρέπει να συμμετέχουν σε εκστρατείες συνειδητοποίηση και πολιτικές. Υπάρχει και το θέμα ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γυναικών όπως και μεταξύ των ανδρών. Γι' αυτό πρέπει αυτές τις αλλαγές, αυτές τις διαφορές μάλλον, συγγνώμη, αν πρόκειται για νέες γυναίκες, για ηλικιωμένες, αν πρόκειται για γυναίκες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ή που είναι πολύ λιγομορφωμένες, πρέπει να εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο όταν ετοιμάζουμε τις πολιτικές μας. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να φέρουμε και να, όλο και περισσότερο τη συζήτηση για την ε, ισότητα των δύο φύλων στην ε, δημόσια συζήτηση. Είναι σημαντικά θέματα για όλους και για την ανάπτυξη και άρα είναι πολύ σημαντικό το κοινό, η κοινή γνώμη να γνωρίζει τη σημασία που έχει αυτό το ζήτημα. Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που η κρίση το θέμα αυτό το έβαλε στη δεύτερη γραμμή, στα παρασκήνια. Κι όμως είναι πολύ σημαντικό. Και θα έπρεπε να είναι πάνω-πάνω στο κατάλογο των προτεραιοτήτων μας. Τώρα, πώς θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καθορίσουμε ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των δύο φύλων που να συμπεριλαμβάνει όλα τα όργανα, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες που δρούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην είναι μόνο δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα κράτη-μέλη, το καθένα χωριστά. Όχι, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Χρειαζόμαστε έναν καλό συντονιστικό μηχανισμό και σαφή ορισμό του ποιος έχει την ευθύνη γιατί, καθώς και χρονοδιάγραμμα. Τέλος, χρειαζόμαστε και οικονομικούς πόρους και βέβαια σχεδιασμό. Πρέπει επίσης να υπάρχει πιο στενή σχέση με το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και τη στρατηγική για το 2020 μαζί με τις στρατηγικές της διεθνής όπως είναι του Πεκίνου. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή επίσης των χωρών μελών και όπως είπα και πριν όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών για να γίνουμε πιο ισχυροί και να μπορέσουμε έτσι να εφαρμόσουμε τη στρατηγική. Ιδιαίτερα θα έλεγα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε για παράδειγμα να κινητοποιήσουν τις οργανώσεις γυναικών που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν την εφαρμογή της στρατηγικής το ίδιο πρέπει να ζητήσουμε από όλους τους φορείς που δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να υπάρχει δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα ότι θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις αποφάσεις τους. Όλες οι επιτροπές, όλες οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. Πρέπει επίσης, πιστεύω, να υπάρχει μια δεσμευτική ε, απόφαση ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση αυτή του φύλου σε όλες τις διαδικασίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταρχήν και πρέπει και να δημιουργήσουμε και τις ικανότητες ώστε να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά. Άρα χρειάζονται προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό και όλα τα προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό να έχουν και τη διάσταση του φύλου μέσα τους. Συνεπώς το προσωπικό έτσι θα μαθαίνει και θα έχει τα προσόντα για να αντιμετωπίσει σωστά οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διάσταση του φύλου. Πρέπει επίσης να υπάρχει πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους διαφορούς οργανισμούς, η για παράδειγμα, που μπορεί να βοηθήσει με τεχνική αρρωγή και έρευνες. Και αυτό το οποίο κάναμε για να συνοψίσω λιγάκι τι μπορεί να κάνει το κάθε όργανο στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να στηρίζει και η μονάδα για τη διάσταση του φύλου πρέπει να γίνει πιο ισχυρή, με περισσότερους πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομικούς πόρους. Πρέπει να είναι πιο ισχυρή η θέση των μονάδων αυτών στην δομή λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την μνήμα που γίνεται για τη διάσταση των φύλων σε κάθε Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δημιουργήσουμε ίσως μια ειδική μονάδα για τα θέματα ισότητας των φύλων. Ένα τμήμα τέτοιο. Κάθε Γενική Διεύθυνση θα μπορούσε να εκπονεί μία ετήσια έκθεση για το τι πρόοδο πετυχαίνει για την ισότητα των φύλων η κάθε Γενική Διεύθυνση στο δικό της τον τομέα. Και έτσι μετά να έχουμε μία ετήσια έκθεση για την πρόοδο που να επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα και να εντοπίζει την πρόοδο όπου έχει επιτευχθεί για να μπορούμε και να συγκρίνουμε τις γενικές διευθύνσεις, ποιες έχουν προχωρήσει πολύ και ποιες όχι. Και θα έπρεπε να μπορούμε να καταλήγουμε και σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τις χώρες μέλη. Έχουμε και συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να ενισχυθεί η διάσταση του φύλου, να ενισχυθεί ο ρόλος της διάστασης αυτής σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ζητάμε επίσης πιο στενή σχέση ανάμεσα στη στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων και τη στρατηγική 2020. Και ζητάμε η στρατηγική αυτή να αποτελήσει μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να γίνεται και έλεγχος όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και για να ολοκληρώσω για τις χώρες μέλη θα έπρεπε να μας ετοιμάζουν μία ετήσια έκθεση για τη διάσταση του φύλου, όπως κάνουν για άλλα θέματα πολιτικής, να το κάνουν και για τη διάσταση του φύλου και να λένε πώς λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση αυτή στις πολιτικές τους και στη συνέχεια έτσι θα μπορούσαν να είχαν και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τώρα δώσω τον λόγο στους άλλους συναδέλφους, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών της κυρία Στέρ. Καλώς ήρθατε. Και τώρα συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας. Δίνω τον λόγο στην κυρία Μαρία Μαριανόχελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την αξιολόγησή σας. Κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά για την επόμενη έκθεση, την οποία συντάσω ήδη με τη στήριξη των ε, σκιωδών και όλες οι σκέψεις χρειάζονται. Όπως και εσείς είδα βεβαίως τα ισχυρά σημεία της προηγούμενης ε, στρατηγικής που είναι ότι υπάρχουν πέντε τομείς προτεραιότητας Αλλά βεβαίως υπάρχουν και αδυναμίες, ε, δηλαδή η στόχοι αυτοί, τα κονδύλια και όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην στρατηγική. Υπάρχει δηλαδή ελάχιστη εστίαση στην νομική υποχρέωση του τι πρέπει να εφαρμοστεί δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δηλαδή τι γίνεται αν δεν συμβούν τα πράγματα. Επίσης σημαντικό είναι στην ε, επόμενη στρατηγική να τα δούμε αυτά. Το αναφέρατε και εσείς. Ε, να δούμε άλλους τομείς, όπως το περιβάλλον, η κινητικότητα, η φορολογία, μετανάστευση, ΜΜΕ, όλα αυτά να μπουν. Και βεβαίως ε, και η χρηματοδότηση και η στελέχωση πρέπει να αναφερθούν. Από την δική σας την πλευρά αναφέρθηκαν οι άντρες ως ε, ομάδα στόχος, ε, παραδείγματος χάρη στη βία κατά των γυναικών. Γιατί είναι συχνά οι δράστες. Και βεβαίως ε, πρέπει να δούμε πως υπάρχουν και άντρες που ε, μειονεκτούν λόγω του φίλου τους. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Οι άντρες δηλαδή, εντάξει μπορούμε να τους δούμε ως δράστες, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Να μάθουμε επίσης και από τα υφιστάμενα κείμενα. Ποιος κάνει τι και πότε. Αυτή η κατανομή δηλαδή. Ποιος είναι αρμόδιος για τι πράγμα και πότε και με αξιολόγηση νομίζω είναι ε, σημαντικό. Το αναφέρατε και στην ε, τελευταία έκθεση. Η Κομισιόν έχει κάποια πράγματα να κάνει οι γενικές διευθύνσεις, τα κράτη-μέλη και βεβαίως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι αυτό με κάποιες προθεσμίες που θα ελέγχονται. Γιατί ακριβώς το θέμα είναι μια καλή στρατηγική η οποία υπήρχε να εφαρμοστεί. Γιατί αυτό δεν είχε γίνει. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μια όθηση για να επιτύχουμε κάτι για τις γυναίκες επιτόπου. Κρίμα είναι βεβαίως ε, κοιτώντας την παλιά στρατηγική ε, και δεν ξέρω αν έχετε κάποια άποψη αν ε, είχε διαδοθεί καθόλου στη δημοσιότητα. Ήταν εσωτερικό έγγραφο ή βγήκε έξω στους ενώσεις γυναικών, στις κυβερνήσεις. Νομίζω πως αυτό είναι μια σαφής αποστολή της επόμενης στρατηγικής. Δηλαδή η δημοσιότητα να μην περιοριστεί εδώ μέσα αλλά τα 28 κράτη-μέλη να μάθουν ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική, να γίνουν ε, κάποια φυλάδια για τη στρατηγική αυτή, για να τη γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης ε, πρέπει οτιδήποτε βγαίνει από το Κοινοβούλιο να περιέχει αυτό το σχέδιο δράσης. Πολύ ωραία ήταν η απαρίθμησή σας για τις συστάσεις. Το ότι υπάρχει αυτή η ιδέα δηλαδή ότι η πολιτική του φίλου θα πάει σε μια μικρή ομάδα που θα ασχολείται και όλοι οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν τη δουλειά τους βλέπετε ότι έχει αποτύχει χρειάζεται κάποια συνεργασία. Είδατε πως πρέπει να έχουμε αυτή την υποχρεωτική αξιολόγηση αντικτύπου σε όλους τους τομείς της πολιτικής. γιατί υπάρχει παραδείγματο χάρη υποχρεωτική αξιολόγηση αντικτύπου η οικονομική για οποιοδήποτε πολιτικό βήμα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για τον τομέα των γυναικών. Ελπίζω να μου επιτρέπετε να έρθω σε επαφή μαζί σας για τη νέα στρατηγική που καταρτίζουμε. Ήταν πάρα πολύ σωστά αυτά τα οποία είπατε και ήρθαν πραγματικά την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να σας ευχαριστήσω και αναμένω και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ε, ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει. Τον λόγο έχουν οι σκιώδεις Η κυρία Γκάλ Πέλτς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν ξέρω, είναι εδώ. Έχει στείλει κάποιον άλλον. Την αντικαθιστά κάποια. Όχι. Κυρία Βυσνιεύσκα, ούτε αυτή είναι εδώ. Από το ECR όχι. Άλντε, κυρία Μιλίναρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με την εισηγήτριά μας και με τα όσα είπε λεπτομερώς πολύ καλή η εκθεσή σας ε, και η εξηγήσει σας εις βάθος. Και όπως είπε και η συνάδελφος, ε, σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε αυτά στην Επιτροπή. Το βασικό πράγμα που τονίσατε εδώ είναι πως ε, το ζήτημα του φίλου δεν πρέπει να είναι κάτι το απομονωμένο, αλλά κάτι το οποίο θα υπάρχει παντού. Και αυτή είναι και η προσωπική μου προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την Γκουε, η κυρία Μπιόρκ ή κάποιος άλλος. Όχι, δεν είναι εδώ. Μάλιστα, πράσινη. Φαντς τορτας όχι, ούτε αυτός είναι εδώ. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, όχι. Ωραία, κυρία Πέτια τότε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτής της τόσο λεπτομερούς έκθεσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ε, σε ποιο βαθμό και πώς πιστεύετε ότι η πλατφόρμα δράση του Πεκίνου εφαρμόζεται. Δηλαδή τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ε, για αυτή την πλατφόρμα δράση του Πεκίνου, την εφαρμόζουν και σε ποιο βαθμό. Κάτι που για μένα είναι σημαντικό και δεν είναι αρκετά γνωστό στο κοινό είναι ότι σε μια διάσκεψη για την ανάπτυξη και τον ε, πληθυσμό ελέγχθη ότι οι αμβλώσεις δεν θα πρέπει να γίνουν τμήμα του οικογενειακού προγραμματισμού. Ε, θα πρέπει να προλαμβάνονται οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ε, και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να και με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε την ανάγκη ε, των αμπλώσεων. Τα κράτη-μέλη όμως δεν έχουν κάνει και πολλά πράγματα που σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν την εντύπωση. Θα κάνετε κάποια σύσταση για αυτό το ζήτημα. Ίσως δεν είχατε βέβαια πολύ χρόνο, γι' αυτό δεν το αναφέρατε στην εκθέσή σας. Ευχαριστώ. Στο κύριος Ταραμπέλα έχει τώρα το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους συντάκτες της έκθεσης. Ε, μαζί με τους κοιόδης εισηγητές θα έχουμε την ευκαιρία να, σας, να μιλήσουμε ξανά για αυτό το θέμα των εξέλιξεων σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων. Ε, σήμερα ή αύριο δεν είμαι σίγουρος. Ε, η έκθεση λοιπόν αυτή είναι και θα είναι πολύ χρήσιμη. Εστιάζοντας τα δικαιώμα, στο δικαίωμα της ε, γυναίκας ε, να χειρίζεται όπως επιθυμεί το σώμα της και με ελεύθερη πρόσβαση σε αντισυλληπτικά, ε, σε αντισύ, στην αντισύλληψη μάλλον και στις αμβλώσεις, βλέπουμε ότι δυστυχώς η θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες, μέσω σεξουαλικής διαπαιδαγωγής. Βέβαια, όταν μιλάμε για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, οι ίδιοι οι οποίοι ε, οργίζονται με τις αμβλώσεις ε, και θέλουν να τις απαγορεύσουν, ε, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι διαφωνούν με την εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος στα σχολεία. Ορισμένοι και κυρίως άντρες θεωρούν ότι η άμβλωση ε, είναι, είναι μια μέθοδος αντισύλληψης. Όχι, θα πρέπει να προωθήσουμε άλλες μεθόδους αντισύλληψης. Ε, χαίρομαι που ο ίδιος ο Πάπας ε, δεν είναι τόσο απόλυτος στη σκέψη τόσο η προηγούμενη προκατοχή του. Η αντισύλληψη είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δίδεται ενημέρωση. Συνεπώς χωρίς να αρνηθούμε το δικαίωμα στην άμπλωση Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε και τις νέες γυναίκες, τις κοπέλες αλλά και τα αγόρια για τις μεθόδους αντισύλληψης. Ε, είμαστε λίγοι εδώ οι άντρες βέβαια σε αυτή την ε, επιτροπή. Ε, ε, παρόλα αυτά ε, η, η μέρα της Λευκής Κορδέλας είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από άντρες στον Καναδά. Ε, ε πάση περιπτώσει θα πρέπει και εμείς εδώ να επιθυμούμε και να προσπαθούμε όλο και περισσότεροι άντρες ε, να ε, κάνουν δικό τους τον αγώνα για την ισότητα των δικαιωμάτων και να μάχονται στο πλευρό των γυναικών. Μόνο έτσι η κοινωνία η οποία κατά βάση δεσπόζεται από άντρες, την οποία δεσπόζουν άντρες, θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση της ισότητας. Ευχαριστώ. ešte, či sú ďalšie pani pani by Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Όχι. Τον λόγο έχει πάλι η κυρία Σαμακά για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στην διάθεσή σας αν θέλετε κάτι. Γεγονός είναι πως θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών και των άλλων ε, θεσμικών οργάνων για την εφαρμογή της νέας ε, στρατηγικής, ειδικά για τα παιδιά εκείνα στα οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα εμπλοκή. Και τώρα θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η αξιολόγηση αντικτύπου για το φύλλο, προϋπολογισμοί για το φύλλο και πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο για να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Όσον αφορά το θέμα των εκτρώσεων δεν αναφέρεται νομίζω ρητός ε, στην ε, πλατφόρμα. Αυτό το οποίο αναφέρεται είναι το θέμα των ε, γυναικών, της υγείας των γυναικών και αυτό είναι ένας τρόπος όταν παραδείγματος χάρη αφορά τα παιδιά ή τις δυσκολίες που υπάρχουν επίσης ε, σχετίζεται μέσως με τη βία κατά των γυναικών, συχνά, καμιά φορά μάλλον η έκδοση είναι από τα... προέρχεται μετά από μία βία. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, αλλά πρέπει να στηριχθούν. Και βέβαια έχει σχέση και με το ζήτημα της φτώχειας ε, και της γυναίκες στην οικονομία. Π.χ. μπορούμε να στηρίξουμε τις γυναίκες, να, έχουν, να κάνουν παιδιά μαθαίνε, και να μπορούν να τα ταΐσουν, να δουλέψουν άμα θέλουν, γιατί θα υπάρχουν υπηρεσίες να τις στηρίζουν. Πρέπει λοιπόν να το δούμε το ζήτημα ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα είναι η κατάσταση των γυναικών στις ε, χώρες του κόλπου. Παρακαλώ την κυρία Μισελ Αλιο Μαρίνα έρθει εδώ και να αναλάβει την Προεδρία. Buenas Καλησπέρα σα. Ξεκινάμε με το σημείο 5 τη σημερινής διάταξη: η κατάσταση των γυναικών στα κράτη του κόλπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τα άτομα και για την ακρίβεια το άτομο ε, την κυρία Ραχίλ Ροτσάζ, η οποία θα παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Δεν ξέρω αν το πρόφερα καλά. Να καλωσορίσω και τον πρέσβη, που είναι νομίζω παρόν εδώ. Δίνω μέσω στο λόγο στην ε, πρόεδρο της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις ε, χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, την κυρία Λιωμαρή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή σας και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Χαίρομαι που λαμβάνει η χώρα η σημερινή συνάντηση. Πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος να εργαζόμαστε. Να μην εργάζεται ο καθένας ε, στη δική του αντιπροσωπεία η Επιτροπή, αντιθέτως να προσπαθούμε πάντοτε να αποκτούμε μια πιο οριζόντια και σφαιρική άποψη των πραγμάτων. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ε, και για το οποίο θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση της κυρίας Ρότσας είναι ένα πραγματικά καλό παράδειγμα γιατί στην δική σας επιτροπή ε, επεξεργάζεται θέματα σχετικά με τις γυναίκες ε, στην δική μας αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του κόλπου ε, ασχολούμαστε με θέματα οικονομικά, πολιτικά αλλά και ανθρώπινα, ανθρωπιστικά ε, που άπτονται αυτής της περιοχής. Ως ε, πρώην Υπουργός Άμυνας ε, έχω επισκεφθεί επανειλημμένως τις ε, περιοχές του κόλπου, χώρες του κόλπου ε, και με έκπληξη είδα σε κάποια λίγα ελάχιστα χρόνια από το 2002 και μετά ε, να έχει καταγραφεί σημαντική εξέλιξη σε ορισμένε χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Οι, οι χώρες του κόλπου έχουν υπογράψει την Σύμβαση για την κατάρριξη των διακρίσεων των γυναικών όλες οι χώρες του κόλπου την έχουν επικυρώσει. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια εκρεμή θέματα. Βλέπουμε βέβαια γυναίκες πολιτικούς, κάτι το οποίο ήταν ε, άγνωστο παλιότερα. Ε, όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των γυναικών. Σε ορισμένες χώρες ε, δίδεται πολύ σημασία στην εκπαίδευση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κοπέλες ε, πηγαίνουν σχολείο. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες ορισμένων χωρών θα πρέπει να αντιληφθούν το πώς οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη αλλά και στην ασφάλεια και την σταθερότητα των χωρών τους. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την ευαισθητοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2011 υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τις ε, σχέσεις με τις χώρες του κόλπου υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν για να καταπολεμηθεί η βία εναντίον των γυναικών ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνά βέβαια τις ε, χώρες του κόλπου που όμως εκεί και εκεί παραμένει πρόβλημα. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να κάνουμε και προτάσεις έτσι ώστε πρώτον να πετύχουμε αυτή την ευαισθητοποίηση αλλά και δεύτερον να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Η σημερινή συνεδρίαση πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα σημείο κίνησης, ε, θα είναι ενδιαφέρουσα για όλους μας και όλες μας ε, και ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή σας και για την πρωτοβουλία σας η κυρία ρώτησα. Ελπίζω ότι με την παρουσία τη θα μα επιτρέψει να δούμε το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βάθο. Yes. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Τι ε, Τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ τους διοργανωτές μου. Δεν την ευκαιρία να κάνω μια σύντομη παρουσίαση της μελέτης της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών στις χώρες του κόλπου. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε θα περάσω αμέσως στο θέμα μας. Οι χώρες ε, είναι Μπαχρέιν, Ιράν, Ιράκ, ε, Κουβέιτ, ε, Ομάν, Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλφαβητικά στο λατινικό αλφάβητο όλες οι χώρες που βλέπετε δηλαδή στο χάρτη εκτός από την Ιεμένη. Βεβαίω η περιοχή είναι γνωστή για τον πλούτο της, τον πετρελαϊκό και άρα έχει σημαντική πολιτική και οικονομική επιρροή παγκοσμίω και στο τοπικό επίπεδο. Επίσης ε, προφανώς είναι μια μουσουλμανική περιοχή και είχε και αρκετούς πολέμους ε, προσφάτως αλλά και στο παρελθόν. Αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό όμως είναι η ανομοιογένεια της ιστορικής ε, πορείας, η εθνοτική ποικιλομορφία, οι διαφορές όσον αφορά επίσης ε, τον πληθυσμό και ο αριθμός των μεταναστών στις διάφορες χώρες. Να δούμε τώρα τη διαφορετική ιστορία της ε, κάθε χώρας. Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το πεδίο αυτής της μελέτης. Αλλά σημαντικό είναι πως ε, υπάρχουν εκεί πέρα Άραβες, ε, Αρμένοι, Βαλούχοι, Κούρδοι, ε, Πέρσες βεβαίως και Τούρκοι. Ειδικά το Ιράν είναι πολυεθνική κοινωνία και υπάρχουν βουδιστές, σιήτες, σιήχες, σιήτες Σουνίτες, ε, Χριστιανοί και Εβραίοι. Σημαντικός είναι ο αριθμός των μεταναστών. Το ποσοστό κυμαίνεται από κάτω από 1% στο Ιράκ μέχρι 70% του πληθυσμού του Κατάρ που είναι μετανάστες. Ε, εδώ πέρα ε, ζόμαστε κυρίως και εν μέρη στην κατάσταση των γυναικών μεταναστών. Παρατηρούν πως κάποιες χώρες έχουν νόμους για να προστατεύουν τους ε, μετανάστες ε, που άλλες φορές περιλαμβάνουν και άλλες φορές όχι τους, ε, τις οικιακές βοηθούς. Συχνά δεν ξέρουμε αν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι και αν οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Οπότε δεν έχουμε πληροφορίες. Για το λόγο αυτό χρειάζεται περισσότερο έρευνα ακριβώ για αυτέ τι ε, ομάδε, ε, τι γυναίκε δηλαδή, μετανάστες. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι πω τα τελευταία 30 χρόνια η περιοχή έχει παγκοσμιοποιηθεί, ειδικά από την τεχνολογική σκοπιά. Η διαδικασία αυτή σημαίνει πως ε, κάποια πολιτισμικά, θρησκευτικά και πολιτικά όρια τονίζονται, παραδείγματος χάρη μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, των φυλών και των αστικών περιοχών και Αράβων και λοιπόν. Και αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη όταν αναλύουμε την κατάσταση των γυναικών καθώς το φύλλο και η σεξουαλικότητα είναι ζητήματα που αποτελούν ε, ακριβώ ε, ένα σημείο οριοθέτησης μεταξύ των ομάδων. Εδώ λοιπόν ε, υπάρχει η πολιτική λεγόμενη της ταυτότητας και αυτό σημαίνει πως οι προσπάθειες διεθνών δυτικών οργανισμών μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν ένα χαρακτήρα οριενταλιστικό, απεικιοκρατικό, πατερναλιστικό, οπότε είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα της συνεργασίας για τα θέματα γυναικών. Οπότε η εργασία πάνω σε αυτά τα ζητήματα θεωρείται μια πολιτιστική εισβολή της δύση και μπορούμε να πούμε πως τα αντιδυτικά αισθήματα είναι αρκετά διαδεδομένα και μεταξύ των γυναικείων οργανώσεων και ακτιβιστών της περιοχής. Η Σαρία είναι το βασικό νομικό πλαίσιο για τις χώρες αυτές. Είναι βάση των νομοθετικών συστημάτων, όμως όλες αυτές οι χώρες έχουν μεικτά συστήματα. Ασίζονται στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, το αγγλικό αστικό δίκαιο, το γαλλικό αστικό δίκαιο, το αιγυπτιακό δίκαιο, εθιμικό δίκαιο κτλ. Στα συντάγματα αυτών των χωρών, τα αστικά δικαιώματα των πολιτών αναγνωρίζονται εξαρτήτως ε, καταγωγής και θρησκείας, όμως η Σαρία είναι το γενικό πλαίσιο που καθορίζει το εάν κάτι επιτρέπεται ή όχι. Και αυτό σημαίνει πως για τα θέματα εκείνα τα οποία δεν καθορίζονται ρητός στο Σύνταγμα, οι δικαστές ε, έχουν την εξουσία να βασιστούν ε, στο πώς ερμηνεύουν οι ίδιοι την Σάρια. Και βεβαίως έτσι το σύστημα καθίσταται αφέρετο και δεν υπάρχει μια εγγυημένη εφαρμογή αστικών δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών. Υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους ε, οι νόμοι των οχτώ χωρών που μας ενδιαφέρουν ε, ομοιάζουν. Π.χ. στο δικαίωμα επιμέλειας του παιδιού, διαζυγίου, ελευθερίας ταξιδίου, βλέπουμε πως υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Υπάρχουν περιορισμένοι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται να ζητήσουν διαζύγιο οι γυναίκες, ενώ οι άντρες μπορούν να ζητήσουν διαζύγιο μόνο μερός. Οι γυναίκες μπορούν να ζητήσουν διαζύγιο βεβαίως και αυτές μόνες τους, αλλά αυτό σημαίνει πως χάνουν τα δικαιώματα που αναφέρει η ε, σύμβαση που υπέγραψαν με το γάμο. Την πρίκα τους δηλαδή πρακτικά. Όσον αφορά την επιμέλεια, μέχρι μία ηλικία παίρνουν το, τα παιδιά γυναίκες και μετά εξαρτάται ε, από την κάθε χώρα. Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν αν θα πάνε με τον πατέρα ή τη μητέρα τους. Όμως ε, ε, οι πατεράδες παραμένουν και οι δαιμόνες. Οπότε αποφασίζουν τα σημαντικά ζητήματα. Εκπαίδευση, ταξίδια, ιατρική φροντίδα κτλ σε πολλές χώρες οι γυναίκες δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς την γυναίκα του και δαιμόνα τους, πατέρα ή συζύγου, ειδικά αν θέλουν να φύγουν από τη χώρα και ακόμα και στις χώρες που δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όπου μπορούν να ταξιδέψουν οι γυναίκες, υπάρχουν ακόμα κάποιοι κοινωνικοί περιορισμοί που ίσως τις αποτρέπουν. Όσον αφορά τώρα τα θέματα κληρονομιάς ή την αποζημίωση για δολοφονία κάποιου συγγενούς και την κατάθεση επίσης ε, στα δικαστήρια. Σε όλα αυτά η γυναίκα αξίζει το μισό από τον άντρα. Είτε μιλάμε για κληρονομιά, είτε για αποζημίωση, αλλά ακόμα και στο δικαστήριο η ε, μαρτυρία της γυναίκας έχει τη μισή αξία της μαρτυρίας του άντρα ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Η βία κατά των γυναικών συγκεκριμένα ε, δεν ε, αναφέρεται στους νόμους. Εμπίπτει σε ένα γενικό πλαίσιο σωματικής προστασίας των πολιτών. Αλλά βλέπουμε στις συγκεκριμένες εκθέσεις μας σαν χώρα πως θέλουν οι αρχές ε, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών και να αναλύσουν επίσης ε, ε, το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο που διευκολύνει τη βία. Τέλος, ε, τέλος εννοώ για αυτή τη διαφάνεια, τα ζυγάρια μπορούν στα προγαμιαία συμβόλαιά τους να ορίσουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Αλλά βεβαίω αυτό είναι θέμα συνεννόηση μεταξύ των συζύγων και τη σημασία που αποδίδουν στην ισότητα των γυναικών. So, um, did I miss one? In the next uh, diagram, I'd like to... Το επόμενο διάγραμμα τώρα θα ήθελα να σας δώσω κάποιες στατιστικές πληροφορίες για την οικονομική συμμετοχή των γυναικών, τα στοιχεία του 2012. Το κόκκινο είναι ποσοστό που απασχολείται σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δηλαδή αμοιβόμενη εργασία από μια ηλικία νόμιμη και πάνω. Το μαύρο χρώμα είναι ανέργειες, δηλαδή γυναίκες που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. Το πράσινο είναι εκτός ε, της εργασίας. Δηλαδή δεν θέλουν και δεν έχουν δουλειά. Βλέπετε τεράστιες διαφορές. Αν συγκρίνετε παραδείγματος χάρη το Ιράκ με το Κατάρ. Και βεβαίως η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή πρόκειται για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο και στο Υπουργικό Συμβούλιο. βλέπουμε εδώ πέρα το Ιράκ που έχει 82 βουλευτίνες. Αυτό είναι, το έχει καταφέρει χάρη σε μια ποσόστοση. Αλλά βεβαίω δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά τις υπουργούς. Επίσης οι, πολιτικοί, οι γυναίκες πολιτικοί στο Ιράκ αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ασφάλειας καθώς παρενοχλούνται μόνο και μόνο επειδή είναι πολιτική, κάτι το οποίο θεωρείται μη πρέπον ως ένα βαθμό. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε τον αριθμό των γυναικών στο Σαουδαραβικό Κοινοβούλιο, αλλά είναι κάπως περίπλοκο το πολιτικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας με την έννοια ότι ο βασιλιάς και η βασιλική οικογένεια έχουν τεράστια εξουσία και υπάρχουν απλά κάποια συμβουλευτικά σώματα και τοπικές συνελεύσεις ε, στα οποία συμμετέχουν οι γυναίκες ε, αλλά δεν είναι σαφές ε, το εάν έχουν πραγματική εξουσία οι γυναίκες ή όχι. Επιπλέον οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία διορίζονται από την βασιλική οικογένεια, κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, όταν φτάσουν σε μια τέτοια θέση αυτό σημαίνει πάντα με τρόπο ελεγχόμενο. Ο αριθμός ε, των ε, γυναικών υπουργών σε όλες τις χώρες είναι χαμηλός. Κάπως διαφέρει η κατάσταση στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως στο Μπαχρέιν οι διασυνδέσεις με τη βασιλική οικογένεια είναι σημαντικές για να θεωρηθεί κανείς ε, κατάλληλος για θέσεις εξουσίας. Και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα οι γυναίκες ε, που είναι γνωστές έχουν πρόσβαση και σε ε, πολιτικές θέσεις. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο το γενικότερο για να αντιληφθούμε το τι σημαίνουν. Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα πράγματα είναι κάπως καλά στις χώρες του κόλπου. Βλέπουμε τον υψηλό αριθμό γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστημιακό πτυχίο και πάνω. Δυστυχώς στοιχεία για το Ιράκ δεν έχουμε, λόγω της ε, κατάστασης των τελευταίων ετών. Ε, και δεν, υπάρχει, βεβαίω, ε, δεν υπάρχουν οι συνθήκες για έρευνα, ούτε για αυτό το ζήτημα, ούτε για άλλα. Το διάγραμμα δείχνει το ποσοστό γυναικών και ανδρών που έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές και ανώτερες σπουδές από την ηλικία των 25 και πάνω. Ε, δυστυχώς ε, οι χρονιές δεν είναι όλες οι ίδιες για όλες τις χώρες, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Από την άλλη, ένα υψηλό ποσοστό εκπαιδευμένων γυναικών εξηγείται και από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για σπουδές στο εξωτερικό τις οποίες εκμεταλλεύονται κυρίως οι άντρες γιατί οι ανήπαντρες γυναίκες ε, έχουν λιγότερες πιθανότητες να πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν χωρίς την οικογένειά τους τα νούμερα αυτά περιλαμβάνουν μόνο όσες ε, ζουν στις χώρες αυτές ε, τη στιγμή της έρευνας. Με βάση λοιπόν τα ευρήματά μας κάνουμε κάποιες συστάσεις. που θα έπρεπε να σκεφτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις τους με τις χώρες αυτές για να ενισχύσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Θα αναφέρω λίγα πράγματα χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Πιο πλήρη στοιχεία βλέπετε στο κεφάλαιο 6. Πρώτον, να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων. Μιλάμε για συμβάσεις που έχουν κυρωθεί όπως η ΣΥΝΤΑΡ το Ιράκ είναι η μόνη χώρα που δεν την έχει κυρώσει. Κάποιες χώρες του κόλπου ε, θεωρούν πως η σύμβαση αυτή δεν συμβιβάζεται με την Σαρία. Ε, υπάρχουν όμως γειτονικέ μουσουλμανικές χώρες που την έχουν ήδη εφαρμόσει. Ε, μπορούμε να διευκολύνουμε κάποιες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να οργανωθεί ένας διάλογος μεταξύ εκπροσώπων αυτών των χωρών για να υπάρξει μια ανταλλαγή ιδεών για το πώς η σύμβαση αυτή σύντομα θα μπορέσει να συμβιβαστεί με τη Σαρία. Κατόπιν έχουμε μια ενσωμάτωση στρατηγικής του φύλου στην σχετική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βεβαίως θα δείτε στο κεφάλαιο 5, τα προγράμματα αυτά είναι περιορισμένα παρά το ότι το Εράσμος παραδείγματο χάρη έχει ως στόχο την ισότητα. Μπορούσαμε να αναλύσουμε εάν ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Εράσμους ε, ωφελούν εξίσου άνδρες και γυναίκες. Κατόπιν, η προώθηση ακαδημαϊκών ανταλλαγών και η συνεργασία στην διεθνή έρευνα για τα ζητήματα του φύλου, κάπως ήπιο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραδείγματος χάρη για το Ιράν, καθώς οι σχέσεις με τη χώρα αυτή είναι πολύ περιορισμένες. Επίσης να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των γυναικών στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τις θεωρήσεις. Αυτά είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές και ήδη υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά τα δικαιώματα των γυναικών θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα. Τέλος, να στηριχθούν γυναικείες ΜΚΟ και γυναίκες πολιτικοί. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ε, δυτική παρέμβαση στα εσωτερικά των χωρών αυτών και να έχει και αρνητικές συνέπειες για τους ενδιαφέρομε τις ενδιαφερόμενες πολιτικούς και ΜΚΟ. Οπότε πρέπει να το δούμε προσεκτικά ασχοληθούμε με κάπως ε, πιο ακίνδυνους ε, τομείς όπως η καταπολέμηση της φίας κατά των γυναικών. Τελευταία διαφάνεια λοιπόν αυτή. Είχαμε διάφορους ερευνητές. Υπήρξε και Υπήρξαν και κάποιοι που έλεγξαν μετά την έκθεση αυτή, την αναθεώρησαν, αλλά δεν θα αναφέρω τώρα τα ονόματα. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, ερευνητέ οι οποίοι ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Το λόγο τώρα έχει ο πρέσβης ο κύριος Χαμίτ Σαλέ Μασούρη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πρέσβης των Ηνωμένων Εμμυράτων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Πρόεδρε και εσάς που παρουσιάσατε την ε, εισήγηση αυτή και σας ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέψατε να έρθω και να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία ενημερωμένα για την κατάσταση ιδιαίτερα στη χώρα μου, στην Ομένα Εμμυράτα και ιδιαίτερα μάλιστα εκεί. Ε. Όπως αναφέρονται και τα στοιχεία στην έκθεση, πρόκειται για το 2002 ή 2008, ενώ τώρα είμαστε σχεδόν στο 2015. Τα τελευταία 43 χρόνια τα Ηνωμένα Μοιράτα έχουν ε, προχωρήσει πάρα πολύ. Αύριο μάλιστα έχουμε την εθνική μας ε, γιορτή, 43η. Έχει γίνει πρόοδο στην οικονομία, την εκπαίδευση, στην πολιτική, στα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά άλλα. Συνεπώς η νομοθεσία έχει επίσης προσαρμοστεί για να είναι προσαρμοσμένη με τις διεθνείς προδιαγραφές. Δημογραφικά η χώρα μας έχει μια ιδιαίτερη δομή. 80% βρίσκονται εκτός της χώρας. Συνήθως που ουσιαστικά το 80% είναι μετανάστες μάλλον που ζουν στη χώρα και μόνο το 20% είναι ντόπιοι. Και στέλνουν χρήματα σε πολλές και διάφορες χώρες όλοι αυτοί οι μετανάστες όπως καταλαβαίνετε. 9 εκατομμύρια. Είμαστε με 1 εκατομμύριο ντόπιου και 8 εκατομμύρια μετανάστες. Θέλω να διευκρινίσω δύο σημεία στην παρουσίασή σας. Το 41229 που αναφέρεται στις εθνικές μειονότητες και τις διεθνείς σχέσεις. Ότι ένα παιδί από γυναίκα από τα Ηνωμένα Εμμυράτα αλλά πατέρα από το εξωτερικό δεν μπορεί να έχει την εθνικότητα της χώρας. Δεν είναι αλήθεια. Το 2012 υπήρξε νόμος που λέει ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί ένα παιδί να ζητήσει την υπηκότητα. Και αυτό ισχύει τώρα στην πράξη. Στο 14.2.2.10 οι μετανάστριες, το εργατικό δυναμικό. Λέτε ότι δεν αναγνωρίζονται ως μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας και άρα αποκλείονται από προστασία το οποίο όμως δεν ισχύει. Πρόκειται για τις οικιακές βοηθούς. Αυτό δεν ισχύει. Γίνεται έλεγχος ακούστηκε ότι γίνονται καταχρήσεις, τους παίρνουν τα διαβατήρια, οι εργοδότες κλπ. Αυτό θέλω όμως να το διευκρινίσω και να πω ότι όλες οι μετανάστριες, είτε είναι και εκεί βοηθοί, είτε δουλεύουν στο εμπόριο, θεωρούνται μέρος του εργατικού δυναμικού μας. Και πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως έρχονται και έχουν σχέσεις με τον εργοδότη με κανονικά συμβόλαια. Δεν είναι ευκαιριακές οι σχέσεις αυτές. Υπάρχουν διάφορες συμβάσει ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων και έχουμε πέρασει πάρα πολλούς νόμους για να προστατεύουμε τους εργαζόμενους και στον τομέα της πρόληψης και της πληρωμής και της κατοικίας και της υγείας. Ένα από τα μέτρα που ισχύει ρυθμίζει τη σχέση ανάμεσα στις βοηθούς και τον εργοδότη τους. Και η σύμβαση αυτή μιλάει για το δικαίωμα που έχουν και οι δύο πλευρές όσον αφορά τις ώρες εργασίας και ο εργοδότης αναλαμβάνει γενικά όλα τα έξοδα προκειμένου να διασφαλίσει και το, και το κόστος του ταξιδιού της γυναίκας που θα έρθει για να δουλέψει εκεί και καλύπτει την κατοικία κτλ. Το θέμα τώρα της περίθαλψης επίσης είναι κάτι που υποχρεωτικά αναλαμβάνει ο εργοδότης. Οι οικιακοί βοηθοί επίσης έχουν και νομική προστασία βάσει ενός νόμου σταστικό δίκαιο αλλά και του ποινικού δικαίου για να αντιμετωπίσετε το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένα ομοσποδιακό κράτος που αποτελείται από 7 μοιράτα, σαν πρόκειται για 7 κρατήρια. Υπάρχει λοιπόν μια ομοσπονδική κυβέρνηση η οποία καλύπτει όλη την νομοθεσία που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Και το κάθε μοιράτο από τη δικιά του την πλευρά έχει τις τοπικές αρχές που επίσης μπορούν να έχουν λόγο όσον αφορά το εργατικό δυναμικό που κατοικεί εκεί. Εν κατακλείδη λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν τομέα πάνω στον οποίο συνεχίζουμε να δουλεύουμε και γι' αυτό και τα Ηνωμένα Εμμυράτα έχουν δεσμευτεί για να ενισχύσουν όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως. Είμαστε μια από τις πιο δυναμικές χώρες στον αραβικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πάνω από το 70% των αποφύτων όπως είπατε κι εσείς και είναι και σε Υπουργεία, στο Κοινοβούλιο, σε οργανώσεις κυβερνητικές. πιλότοι και συμμετέχουν ενεργά. Και εδώ βλέπετε γύρω μου στην πρεσβεία έχουμε γυναίκες. Τις βλέπετε. Με, μας βοηθούν στη δουλειά, δουλεύουν και εκείνες εκεί όπως και οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Τώρα, συζήτηση. Δίνουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές. Αν κάποιος θέλει το λόγο να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. Όχι. Τότε, Α, παρακαλώ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για τις εμπεριστατωμένες και αναλυτικές ε, εισηγήσεις, ενημερώσεις ως προς το νομικό καθεστώς που υπάρχει. Ε, αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι αν έχει γίνει μια στατιστική καταμέτρηση σε ποιες από τις χώρες στα Εμμυράτα ε, υπάρχει εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας γιατί από αυτά που ακούσαμε σε επίπεδο πληροφόρησης η νομοθεσία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά εκεί που ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα, και αυτό ήθελα να ρωτήσω, είναι στην εφαρμογή του νόμου. Ευχαριστώ πολύ. Sí, la Παρακαλώ κύριε Βαϊνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για τη μελέτη. Μια πάρα πολύ καλή εικόνα και ένα χρήσιμο εργαλείο. Και βεβαίως όπως υπόθηκε έχει σημασία για μας η ισότητα των γυναικών. Τώρα για την σύμβαση ΣΥΔΟ την οποία ε, έχουν ε, συνυπογράψει όλες αυτές οι χώρες ε, εκτός από το Ιράν που θεωρεί πως δεν συμβιβάζεται με την Σαρία, ειδικά το άρθρο 1. Όλες οι υπόλοιπες νομίζω έχουν υπογράψει, νομίζω. Αλλά δεν έχουν υπογράψει το επιπρόσθετο πρωτόκολλο που αφορά την εφαρμογή. Και το τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες σε περιπτώσεις ε, διακρίσεων κτλ. Τι, ε, ποιος έχει λοιπόν η κατάσταση όσον αφορά αυτήν την ε, σύμβαση μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα για να πατήσουν οι ακτιβίστριες για να διεκδικήσουν την ε, ισότητα. Και επίσης σημασία έχει εδώ πέρα, σημασία έχουν και τα στατιστικά στοιχεία για να υπάρχει έλεγχος και μετά εφαρμογή. Γιατί είπατε πως ε, στις περισσότερες χώρες εφαρμόζεται αυτή η συνθήκη. Εδώ πέρα αναρωτιέμαι λοιπόν τι εννοείται ακριβώς ε, εφαρμογή. Γιατί αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε νομίζω απέχουν πολύ ως πραγματικότητα από αυτά τα οποία ορίζει αυτή η σύμβαση. Σας ευχαριστώ. Για να τελειώσουμε, ο κύριος Καν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία πρόσφατα να επισκεφθώ και τον Μπαχρέν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και προσωπικά εντυπωσιάστηκα με τις δραστηριότητες ε, των γυναικών που είδα σε αυτές τις ε, χώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Πολιτικής ε, που κατά βάση ήταν μόνο γυναίκες και αναρωτιέμαι γιατί δεν τις ε, καλέσαμε εδώ πέρα γιατί η συζήτηση αυτή αφορούσε τα ζητήματα ασφαλείας ε, τα οποία και εδώ πέρα βεβαίως απασχολούν κυρίως τους άντρες και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά. Ένα άλλο θέμα είναι το Μπαχρέιν. Χτες είχε τον ε, δεύτερο γύρο εκλογών και υπήρχε αυξημένη συμμετοχή των ε, γυναικών. Αναγνωρίζω βεβαίως ε, την ευαισθησία την οποία αναφέρατε, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ πως αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι πώς θα διαχωρίσουμε κάποιες από τις πολιτισμικές και θρησκευτικές πτυχές αν δείτε προσεκτικά τις θρησκευτικέ πτυχές, ε, νομίζω πως ε, ε, υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός προστασίας από τις πολιτισμικές. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες για να γίνουν αυτές οι αλλαγές τις οποίες όλοι επιθυμούμε για να συνεισφέρουν και οι γυναίκες, κάτι το οποίο πράγματι θα κάνει την διαφορά και νομίζω έτσι θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο κύριος Αλεξανδρίδης έχει το λόγο. Good afternoon. Thank you very much. Καλησπέρα σας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστούμε πολύ το ινστιτουτο ΑΤΡΙΑ για όλη αυτή την έρευνα και την έκθεση των 118 σελίδων. Είναι πολύ ρεαλιστική, βασίζεται σε στοιχεία, δίνει πολλές πληροφορίες. Θα ήθελα απλώς να κάνω μία κριτική. Θα θέλαμε να είχε συμπεριληφθεί και η ΕΜΕΝ γιατί πρόκειται ε, για ε, κρίσιμη χώρα στην περιοχή. Και δεύτερον, θα θέλαμε να είχε υπογραμμιστεί και η απειλή του Ισλαμικού στρατού που βέβαια προσθέθηκε αργότερα στην εικόνα ε, είδαμε όμως ότι στο Ιράκ αλλά και στη Συρία η δράση του Ισλαμικού στρατού ε, οδήγησε σε σημαντικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων γυναικών. Όλα όσα αναφέρεται τα αναφέρουμε και εμείς στις καταχώρα ε, κατά στρατηγικές ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα φύλου αναλύονται αλλά δεν θα πρέπει και να κατακαιρματίζονται. Θα πρέπει να τα βλέπουμε σε ένα συνολικό κοινωνικό πλαίσιο και στο πλαίσιο βέβαια και όλων των υπολείπων δικαιωμάτων. Πολιστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών κλπ. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα δικαιώματα των γυναικών αν δεν ε, εξετάσουμε το αν υπάρχει ελευθερία ε, πίστης, θρησκεύματος, ε, αν υπάρχει ε, θανατική ποινή, Κυρία Τζαμπάρη, για παράδειγμα, η περίπτωση Τζαμπάρη που εκτελέστηκε στο Ιράν ε, επειδή διαμαρτυρήθηκε ότι της ε, επιτέθηκε ε, σεξουαλικά το θύμα. Αυτό δηλαδή, δηλαδή, το θέμα των δικαιωμάτων γυναικών μπαίνει ως εντάσσεται σε όλες τις άλλες πολιτικές Έχουμε πολιτικό διάλογο με τις χώρες του κόλπου, με, την, με το Συμβούλιο των Χωρών του Κόλπου, όχι με όλες τις χώρες ξεχωριστά. Εκεί συζητάμε και θέματα φύλου. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει ε, υπογράψει, επικυρώσει ε, την σύμβαση. Ε, εμείς την οφούμε να το κάνει χωρίς επιφυλάξη, γιατί είναι σημαντικό το θέμα των επιφυλάξεων. Χαίρομαι που που είναι εδώ ο πρέσβης των Ηνωμένων Εμμυράτων με τα Ηνωμένα Αμερικά Εμμυράτα. Έχουμε ένα άτυπο ε, διάλογο για θέματα γυναικών. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στις 20 Νοεμβρίου. Ε, έχουμε καταγράψει σημαντική πρόοδο, πολύ σοβαρή πρόοδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να βρίσκουμε απλώς τα κακά κείμενα και να τα υπογραμμίσουμε ή, από την άλλη μεριά, αυτό που έχουμε εμείς επιλέξει, να υπογραμμίζουμε πάντοτε την πρόοδο ε, και να τη χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα και υπόδειγμα. Ψυχολογικά λειτουργεί καλύτερα γιατί έτσι οθεί και τους γείτονες ε, να ανταγωνίζονται στο ποιος θα πάει πιο μακριά και νομίζω ότι και το, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Θα χρησιμοποιήσουμε την ε, μελέτη αυτή και για το δικό μας προβληματισμό. Ε, γίνεται και μια σύσταση για χρηματοδότηση. Δυστυχώς ο συνάδελφός μου από την ΤΕΒΚΟ δεν είναι εδώ, αλλά γνωρίζω ότι ο καινούριο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, δηλαδή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας, ε, λαμβάνει υπόψη το φύλλο σε μεγάλο βαθμό και είμαι σίγουρος ότι θα δίδει τη δυνατότητα χρηματοδότησης οργανώσεων ε, στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη μελέτη. Ευχαριστώ. Για να τελειώσουμε αυτό το θέμα της ημερησίας ε, διάταξης, δεδομένου ότι ετέθησαν και κάποιες ε, ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Ρότσαρτ. Ευχαριστώ πολύ ε, για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν τις ερωτήσεις του, το θέμα του που έθεσε ο κ. Μασούτη. Ε, δύο σημεία της έκθεσης και είπατε ότι οι πηγές μας δεν είναι πρόσφατες. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε όσο πιο πρόσφατες πηγές γινόταν. Είπατε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ό,τι αφορά την υπηκότητα και την, το, την, νομικό στάτους ε, των οικιακών βοηθών. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Νομίζω όμως ότι ακόμα και έτσι είναι σημαντικό να δούμε και να δείτε το κατά πόσον οι νόμοι αυτοί εφαρμόζονται σωστά. για το, επίσης για το κατά πόσον οι οικιακές βοηθοί γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα επικαλούνται. Σε ό,τι αφορά τις θετικές εξελίξεις, είναι πολύ καλά, πολύ ευχάριστα νέα. Το αναφέραμε μάλιστα ε, στην συνολική μας έκθεση, ίσως όχι τόσο πολύ ε, λεπτομερώς στην καταχώρα ανάλυση, αλλά στη συνολική μας έκθεση το έχουμε πει. Μετά, το θέμα για την διαφορά ανάμεσα στον νόμο, δεν θυμάμαι ποιος έθεσε το ερώτημα, στον το νόμο, οι νόμοι που είναι παρόμοιοι με αυτούς στην Ευρώπη. Νομίζω δικιό σας ερώτημα είναι έτσι. Ε, και για το κατά πόσον εφαρμόζονται σωστά ή όχι. Κατά πόσον έχει, στα, ε, στατιστική, κατά πόσον έχει στατιστικά μετρηθεί αν υπάρχει πράγματι ζήτημα στην εφαρμογή των νόμων. Αυτό, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Όπως το απαντάτε είναι. Το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Yes, exactly. Ναι, έτσι το κατάλαβα. Όχι. Ε, ε δεν έχουμε πληροφορίες για την εφαρμογή. Είναι θέμα περαιτέρω έρευνας. Για το ΣΥΝΤΟ. Ε, για την σύμβαση πράγματι η, η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη που δεν, το έχει, δεν έχει υπογράψει. Όλες οι χώρες έχουν υποβάλει επιφυλάξεις ε, γιατί το θέμα Σαρίας. Η Σαρία δεν συμβαδίζει με την σύμβαση ε, σε όλα τα σημεία. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών, πιστεύω ότι επηρεάζει την κατάσταση των γυναικών Ε, ρωτήσατε αν είναι αξιόπιστο αυτό το πλαίσιο, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Uh, question Η ερώτηση ήταν, πιστεύετε ότι η, σύμβαση αυτή είναι βάση πάνω στην οποία να μπορούν να στηρίξουν τη δράση τους οι φεμιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις των γυναικών. Ε, είναι σημαντική αυτή η σύμβαση για τις οργανώσεις των γυναικών. Ε, ναι, το κατάλαβα. Ω τμήμα τη έρευνά μα, ε, ρωτήσαμε από τους, ε, ζητήσαμε από του εμπειρογνώμονε να μιλήσουν με τι ακτιβίστρε και με τι ε, εκπροσώπου των γυναικών οργανώσεων σε αυτέ τι χώρε. ορισμένοι είπαν ότι θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος εκείνης συζήτηση με των γυναικών. δυστυχώς όμως δεν δόθηκαν τελικά πολλές λεπτομέρειες. Μπορεί να χρησιμεύει αλλά όχι και ιδιαίτερα πολύ αυτή η σήμαση. Σε ό,τι αφορά τη γυναίκες στον Παχρέν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συμφωνώ. Πολύ καλή ιδέα. Ο διαχωρισμός ε, πολιστικών από τα θρησκευτικά ζητήματα, ναι, ε, συμφωνώ. Μία από τις συστάσεις που ανέφερα ήταν να η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές Ισλαμικές χώρες έτσι ώστε να συζητηθεί ακριβώς αυτό το θέμα. Ε, το κατά πόσον η σύμβαση είναι ε, ε, συμβατή με την Σαρία. Ε, ε, η Εμένη, καλό θα ήταν να είχε συμπεριληφθεί βέβαια, ε, αλλά ήδη οκτώ χώρε ήταν αρκετές ε, είπαν οι ερευνητέ, οι επιστήμονε ενδεχομένω σε μια επόμενη μελέτη μα. Muy bien, muchas gracias. Volvo Καλώς. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και συμμετείχατε στην συνάντηση αυτή. Πολύ σημαντική η μελέτη σας και μετά από τη συζήτηση αυτή περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η γνωμοδότηση, η ετήσια γνωμοδότηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο 2013. Η συγκίτρια είναι η κυρία Σινιάνσκα. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τιμή για μένα να μπορώ να σας μιλήσω σήμερα εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βέβαια ζήτημα και όλοι πρέπει τις αξίες αυτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τις προστατεύουμε. Ως συντάκτρια γνωμοδότησης έπρεπε να επιλέξω τα θέματά μου. Ποια θέματα δηλαδή θα συμπεριλάβω στην γνωμοδότησή μου. Είναι ένα περίεργο θέμα. Πάρα πολύ περιπλοκό με διάφορες πτυχές και κοινωνικές ασχολείται με γυναίκες αλλά και άλλες ε, περιθωριοποιημένες ομάδες ε, του πληθυσμού. Όπως ε, είπαμε ήδη η πρόεδρος της Επιτροπής μας λέει πως πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο κρύβεται ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εγώ ασχολούμαι με συγκεκριμένες ιστορίες. Η πρώτη αυτή, η πρώτη ιστορία αφορά μια νεαρή γυναίκα του είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της αφού ε, γεννήθηκαν τα παιδιά της ε, υπήρχε και βία εις βάρος των παιδιών και τελικά η μητέρα αυτή αποφάσισε να τον εγκαταλείψει. αξιέπαινο αυτό, αλλά φοβότανε μην την ξαναβρει και έτσι κρυβότανε σε διάφορους φίλους. Φαντάζεστε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόταν. Οπότε φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Τα είπε και η κυρία Σάμεκ. Και βεβαίως ε, πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και τα προβλήματα των γυναικών. Η έκθεση αφορά και άτομα με αναπηρία, δυστυχώς όμως μόνο σε ένα άρθρο εκεί πέρα που μιλάμε για την ενσωμάτωση της ε, διάστασης ε, του φίλου που λέμε πως θα πρέπει και τα άτομα με αναπηρία να ληφθούν υπόψη και Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χάραξη σωστών πολιτικών χωρίς να συμπεριληφθούν αυτά τα άτομα. Βλέπουμε ε, πως ε, υπάρχει και το σχετικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα το οποίο μας λέει πως συχνά το οποίο μας λέει πως συχνά αγνοούνται και οι αποφάσεις ε, των ε, δικαστηρίων και συχνά υπάρχει πρόβλημα και εμποδίζονται οι γυναίκες με αναπηρία να ξεκινήσουν οικογένεια. Και βεβαίως οι γυναίκες με παιδιά με αναπηρία είναι η πιο ευπαθής ομάδα και θα πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς. Επίσης ε, ένα άλλο θέμα είναι οι γυναίκες σε πολέμους, σε συγκρούσεις, πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα και αυτή για την Επιτροπή μας. Την προηγούμενη εβδομάδα ο, ήρθε και εδώ πέρα ο Δ. Μουκβέγγε για να λάβει το βραβείο Ζαχάροφ και περιέγραψε τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών και θεωρώ πως και η Επιτροπή μας πρέπει να συνεισφέρει έτσι ώστε τέτοιες πράξεις ε, πρέπει να προληφθούν για να μην ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βία κατά των γυναικών στον πόλεμο και πρέπει να τιμωρείται στα δικαστήρια είναι απαράδεκτο και ε, το Τελευταίο θέμα είναι η θέση των γυναικών Ρωμά. Ένα πρόβλημα που είναι γνωστό στις περισσότερες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και υπάρχει και στην Σλοβακία. Γνωρίζω προσωπικά ένα 14χρονο κορίτσι ε, που Ζουν όλοι μαζί, δέκα άτομα σε ένα δωμάτιο, δεν υπάρχει αποχέτευση και η Μαρία, η 14χρονη αυτή, βγαίνει μία μέρα έξω να πάει στην τουαλέτα και τη βιάζουν. Και ήταν, εξάξα να πω ήταν και ανάπηρη. Και Βλέπουμε εδώ πέρα πως οι γυναίκες είναι θύματα της βίας ακόμη μια φορά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη συνθήκη ζωής αυτών των γυναικών, των κοριτσιών, που συχνά φεύγουν και από το σχολείο ή δεν πάνε καν σχολείο, είναι έγκυος πάρα πολύ πάρα πολύ νωρίς και το θεωρούν αυτό μια πηγή εισοδήματος. Γι' αυτό γίνονται μητέρες ε, πολύ νωρίς. Αυτό είναι πρόβλημα της ε, κοινωνίας. Ε, έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός και γνωρίζω πραγματικά εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις και θεωρώ πως θα έπρεπε στο μέλλον να υπάρξει κάποια στήριξη αυτών των γυναικών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας γιατί νομίζω πως ε, έχετε κι εσείς τις ίδιες προτεραιότητες με μένα και θα μπορέσουμε από κοινού να προωθήσουμε αυτές τις εκθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Συνάτσκα για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Συζήτηση τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Πετήρ. Η σκιώδη συγκίτρια, η Μαρία Γκαμπριέλ, μου ζήτησε να παρουσιάσω την ε, αξιολόγηση της έκθεσης αυτής. Θέλει τους χαιρετισμού και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Είναι στο Στρασβούργο σε συνάντηση της Κοινής Κοινοβουλευτικής της Κοινοβουλευτικής ε, Επιτροπής ECI. Θέλω λοιπόν να σας πω τα εξή εκ μέρους της. Πιστεύει ότι το σχέδιο αυτογνωμοδότησης περιλαμβάνει τις παραγράφους 56 έως 61 που αναφέρονται στη βία κατά των γυναικών. Την τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων και άλλα. Θέλω λοιπόν, θέλω λοιπόν ευχαριστήσει την κυρία Σινάντσκα για την έκθεσή της. Πιστεύει όμως ότι θα έπρεπε να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο το ρόλο των γυναικών στη δημοκρατία. Γι' αυτό και προτείνουμε τροπολογίες για να ενισχυθεί έτσι ο ρόλος των γυναικών στην ε, οικοδόμηση ειρήνης και την δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι η διάσταση αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί επαρκώς στο σχέδιο γνωμοδότησης. Οι τροπολογίες μας λοιπόν θα έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα. Την καταπολέμηση δηλαδή του ακροτηριασμού των γενετικών οργάνων και τα άλλα που είπα. Επίσης θα έχουμε και μια τροπολογία για τους γάμους που γίνονται σε πολύ μικρή ηλικία και για την πρόσβαση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και θα έχουν να κάνουμε τον ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση ειρήνης. Είναι στοιχεία τα οποία σε ένα βαθμό αναφέρονται στην γνωμοδότηση, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει με περισσότερες λεπτομέρειες να αναφερόμαστε σε αυτά και να δίνουμε κατευθυντήρες γραμμές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Καλώς, δεν βλέπω να θέλει κανένας άλλος το λόγο. Α, εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την γνωμοδότησή σας. το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη ε, συμπεριλαμβάνει και τις ΛΟΑΕΔ. Νομίζω λοιπόν ότι Πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε ότι δηλαδή πολλά από αυτά που αναφέρεται στην ομοδότηση συνάδουμε με τις δικές μας προτεραιότητες. Θα θέλαμε ίσως κάποιες προσθήκες, να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Εμείς για παράδειγμα θα θέλαμε σαφή μνήα στη σύμβαση ΣΥΝΤΟ. Να λέμε δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συζητηθεί και ότι υπάρχουν ήδη διεθνείς συμβάσεις εδώ και χρόνια. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να περιλαμβάνει η γνωμοδότηση είναι να διευκρινιστεί το θέμα της βίας που έχει να κάνει με τη διάσταση του φύλου. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες, έχει να κάνει γενικότερα με την έκφραση του φύλου. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να προσθέσουμε μια παράγραφα προς αυτή την κατεύθυνση. Και όταν μιλάμε για την ε, βία που έχει να κάνει με τη διάσταση του φίλου σε πολέμους, ο Μουγκβέγγε, ακριβώ την προηγούμενη εβδομάδα το βραβείο Ζαχάροφ αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι θα ήθελε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και ανέφερε διάφορες περιπτώσεις. Μίλησε για τη βία στον πόλεμο και είπα ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό αυτό για τις γυναίκες και αυτό που θα θέλαμε εμείς είναι όχι μόνο να αναφέρονται τα προβλήματα αυτά που εντοπίζουμε αλλά να καλούμε και σε δράση. Να λέμε ποια εργαλεία χρειάζονται για να καταπολεμηθεί η βία αυτή που σχετίζεται με το φύλλο. Θα θέλαμε επίσης τη γνωμοδότηση και μια αμνία για τα δικαιώματα, τα αναπαραγωγικά και την αναπαραγωγική υγεία. Γιατί εξακολουθούν πολλές γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση σε τέτοια δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι και αυτό λοιπόν θα έπρεπε να αναφέρεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Το τελευταίο είναι το εξή. Θα θέλαμε μια πιο πολυτομεακή προσέγγιση, γιατί δεν πρόκειται μόνο για διακρίσεις βάση φύλου, πρόκειται και για άλλες ε, διακρίσεις που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό και θα πρέπει να αναφέρονται επίσης στη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η σκιώδης εισηγήτρια, η κυρία Νουρίτσκες επίσης μας έστειλε τα δικά της τα σημεία, γιατί δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ, μας τα έστειλε. Πάνε προς την γραμμή την ίδια που αναφέρατε κι εσείς. Θα ήθελα λοιπόν στη γνωμοδότηση να συμπεριληφθούν, θέλει μάλλον, τρία σημεία να προσθεθούν στη γνωμοδότηση. Πρώτον, μία στην, ε, στη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης γιατί θεωρεί ότι επήγει η επικύρωση από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για δικαιώματα των γυναικών άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια στη γνωμοδότηση από αυτού. Δεύτερον, όσον αφορά τη χρήση των γυναικών που χρησιμοποιούνται σαν πολεμικό όπλο. Να φροντίσουμε για την πρόληψη και για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση και η επίσημη και η άτυπη. Και το τρίτο που θέλει είναι να αναφέρουμε κάτι για την κατάρτιση όλων των ε, φορέων που ασχολούνται με τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Ότι πρέπει δηλαδή να στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες κατάρτισης που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση και να στηρίξουμε όλες τις υπηρεσίες που δουλεύουν για να βοηθήσουν τις γυναίκες που είναι θύματα βίας, γυναίκες και παιδιά. Αυτά. Τώρα, η ημερομηνία για τροπολογίες. 10 Δεκεμβρίου του 2014 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση. Δεν ξέρω, κυρία Ζινάνσικα, θέλει μήπως να απαντήσει στα σχόλια που ακούστηκαν, στις παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ε, θα βρεθεί μια λύση τελικά με την περαιτέρω συνεργασία και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε εδώ παρούσα την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, του ΕΙΓΕ, την περιμένουμε να καθίσει Ε, Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η διευθύντρια του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φίλων, κυρία Λάγκμπακ, ε, είναι παρούσα εδώ σε αυτή την ε, καινούργια επιτροπή δικαιωμάτων της γυναίκας, σε αυτή τη θητεία εννοώ. Θέλω να την ευχαριστήσω που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας ε, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε στενά γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να βρισκόμαστε, να συνδιαλεγόμαστε. Ήθελα να την ευχαριστήσω πολύ ε, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Έχετε το λόγο. Yes, it is. Ναι, και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνω μια τέτοια πρώτη παρουσίαση στην καινούργια σύνθεση της Επιτροπής αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζουμε το πρόγραμμα εργασίας για τον επόμενο χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο το υιοθέτησε πριν από δύο εβδομάδες. Ε, όταν ολοκληρωθεί το κείμενο θα σας το στείλουμε. Σήμερα θα σας δείξω μερικές διαφάνειες μόνο. Ακούγοντας σήμερα για την πλατφόρμα δράσης του, Πε, Πεκίνου, το θέμα του ακροτηριασμού των ε, οργάνων, τα στατιστικά στοιχεία για, τις, ε, για τη βία εναντίον των γυναικών και των ανδρών βέβαια. Ε, η συμμετοχή των ανδρών σε αυτό τον αγώνα ε, ακούσαμε πολλά λοιπόν πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και για μας και για σας. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ε, ο επόμενος χρόνος θα είναι ε, ο τελευταίος, το τελευταίο έτος του δεύτερου κύκλου ε, του τρίτου μας προγράμματος. Θέλουμε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους να έχουμε εγκαθιδρύσει ισχυρές ε, σχέσεις με την Επιτροπή ΦΑΜ ε, και με οποιασδήποτε, οποιαδήποτε άλλα όργανα τα οποία είναι σημαντικά ε, για θέματα δικαιωμάτων, και δικαιωμάτων γενικών και ισότητας των δύο φύλων. Τώρα, εδώ βλέπετε τις, τους βασικούς άξονες της εργασίας αναφέρεται και στον κανονισμό που είναι η νομική βάση μας, αλλά έτσι κι αλλιώς το βασικό μας καθήκον είναι ε, να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και να αναλύουμε τα στατιστικά και τις ε, πληροφορίες που υπάρχουν για θέματα ισότητας των δύο φύλων, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως από πολιτικούς, αλλά και, από, ε, και σε εθνικό επίπεδο, για να αναλυθεί το τι χρειάζεται ε, να γίνει σε επίπεδο πολιτικής μέτρων, δράσεων αλλά και να βασίζουμε σε αυτά τα στοιχεία ακόμα και τον προϋπολογισμό ο οποίος ε, θα δοθεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Έχουμε έναν ε, ποιοτικό δίκτυ τον οποίο ξεκινήσαμε το 2013 για, την, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Τώρα προετοιμάζουμε και ένα δεύτερο δίκτυ το οποίο θα, τον οποίο θα εγγενιάσουμε του χρόνου. Ο δίκτυς αυτός ε, θα αφορά την βία κατά των γυναικών το θέμα αυτό εκκρεμούσε από τον πρώτο δίκτυ. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε και το, και το χώρο εργασίας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός ε, και η Κομισιόν είπε ε, ότι το mainstreaming αφορά το χώρο Ρωσίας και την εργασία γενικότερα. Ε, επίσης, έχουμε το θέμα της, ε, της βάσης δεδομένων για τους δείκτες του Πεκίνου. Ε, βλέπουμε πώς, ε, πόσοι και πώς συνδέονται με αυτή τη βάση δεδομένων, την οποία εμείς επικαιροποιούμε κάθε 6 μήνες, έτσι ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Ε, ε, εστιαζόμαστε όλο και περισσότερο στην βία που εστιάζεται στο φύλλο, δηλαδή στις γυναίκες κυρίως, Θα σας δείξω τι κάνουμε, ποιες είναι οι μελέτες μας και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, επίσης, έχουμε την πολύ βασική περιοχή του, ε, του mainstreaming, το οποίο ε, έχει σχέση με την ευαισθητοποίηση, με την, τους κατάλ, τα την κατάλληλη χρηματοδότηση κλπ. Θα σας πω τι προετοιμάζουμε τον επόμενο χρόνο. Και βέβαια ε, τα ωφέλη της ισότητας των φύλων. Ε, είναι ένα θέμα παγίδα. Χρειαζόμαστε ε, εργαλεία όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά που να αποδεικνύουν το πόσο σημαντική και ωφέλιμη είναι η ισότητα των φύλων. Για τον επόμενο χρόνο προετοιμάζουμε μια έκθεση για την ε, πλατφόρμα δράσης του ε, Πεκίνου κάτι τη διάρκεια της Λουξεμβουριανής ε, Προεδρίας που έχει επιλέξει τις γυναίκες και, την, ε, και τη, λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την έκθεση θα προσθέσουμε και καινούριου δείκτες και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκεφτόμαστε, συζητάμε να επικαιροποιήσουμε και τη βάση δεδομένων για τις γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων ...τη η βάση θα περάσει πιθανώς σε εμάς. Ε, η μελέτη αυτή θα έχει δείκτες για την κοινωνική εξουσία και άλλους δείκτες. Επίσης προετοιμάζουμε ένα ερευνητικό σημείωμα για μία από τις προεδρίες, πιο συγκεκριμένα την Ολλανδική Προεδρία. Και προγραμματίζουμε και την Σλοβακική Προεδρία. Η Σλοβακική Προεδρία θα επιλέξει την ε, ε, εξέταση, να εξετάσει το τι έχει απογίνει η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου. Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο λοιπόν για να συλλέξουμε τα στοιχεία και να τα παρουσιάσουμε στις κυβερνήσεις. Έχουμε επίσης την έκθεση του Πεκίνου. Ε, ε αναφέρθηκε και σήμερα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στην έκθεση για, το, ε, για την πλατφόρμα του Πεκίνου τα οποία θα τα λάβουμε υπόψη. Η έκθεση αυτή δίνει μια ανασκόπηση όλων των θεμάτων. Αναλύουμε τις τάσεις, τα δεδομένα, τις αλλαγές από το 2007 στο 2012 Ορισμένα στοιχεία αφορούν το 2013 μάλιστα. Είναι μια ε, λεπτομερή σύνοψη, θα λέγαμε, για το τι έχει συμβεί σε καθένα από τις τομείς που καλυπτόταν από το Πεκίνο, την πλατφόρμα του Πεκίνου. Και μετά βλέπετε και τις ε, σχέσεις, τις συνεργασίες τις οποίες θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε τον επόμενο χρόνο, έτσι ώστε ε, να ρέουν οι πληροφορίες. Ε, εδώ ε, είναι ε, όλοι οι διάφοροι τομεί, οι δύο ε, κάτω, τα δύο κάτω τραγουνάκια, η βία και οι ε, ε, τεμνόμενες ανισότητες είναι εκεί που εστιαζόμαστε περισσότερο αυτά τα δύο πράγματα αλληλοτροφοδοτούνται δυστυχώς δυσκολευόμαστε να βρούμε στοιχεία και για τις 28 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουμε συγκρίσιμα ε, δεδομένα. Με όλους αυτούς εδώ που βλέπετε τους φορείς προσπαθούμε να συλλέξουμε και να, στοιχεία και να συνεργαστούμε. Ε, τώρα, ε, βάσει δεδομένων για στατιστικά φύλου. Με όποιον και να μιλάω παίρνω θετικές αντιδράσεις. Μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου θέλουμε να έχουμε ήδη εγγενιάσει τη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα όσα έχουμε εντοπίσει εμείς, ε, όλα τα στοιχεία για την ισότητα των φύλων. Όχι μόνο δείκτες, θα έχουμε την βία των γυναικών, θα έχουμε οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες και βάσει δεδομένων, μικρότερες βάσει δεδομένων που διαθέτουμε και θα αναπτύξουμε και ένα ειδικό λογισμικό έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει την έρευνά του. Ε, θα, ο χρήστης θα ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία με βάση κάποιες μεταβλητές ε, και το σύστημα θα του δίνει αυτόματα πίνακες, ε, σχέδια, σχεδιαγράμματα, ε, γραφικές παραστάσεις και τέτοια. Τώρα, σε ό,τι φορά τη βία, το Διοικητικό Συμβουλίο επικύρωσε το πενταετές μας πρόγραμμα που το σχετικό με αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών είχαμε πιο πολλές ε, εκθέσεις από αυτές, αλλά κρατώ τις πιο σημαντικές. Για παράδειγμα είχαμε το θέμα της, ε, ε, του ακροτηριασμού των γενετικών οργάνων των γυναικών. Πριν από δύο χρόνια κάναμε μια ευρωπαϊκή έρευνα, πανευρωπαϊκή έρευνα για το ζήτημα αυτό. Κατόπιν αιτήματος του, της πρώην Επιτρόπου κυρίας Ρέντινγκ, η μελέτη αυτή ε, ήταν η βάση και για ένα κατοπινό ανακοινωθέν. Ε, τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ε, μία μελέτη για τις κοπέλες που κινδυνεύουν. Ε, από τέτοιου είδου ακροτηριασμό. Οπότε είναι η συνέχεια δηλαδή της προηγούμενης μελέτης. Ποιε είναι οι μελέτες, ε, ποιε είναι, οι μέθοδοι, συγγνώμη, είναι, ποια είναι η κατάσταση, πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις πολιτικές που έχουν ε, ή τις εκστρατείε ευαισθητοποίηση για να μειωθεί, μειωθούν αυτού του είδου οι πράξεις. Μετά, το κόστος της βίας είναι μια ε, μελέτη την οποία ήδη τελειώσαμε, θα τη δημοσιεύσουμε στις 8 Δεκεμβρίου, όχι, στις 10, στις 10 Δεκεμβρίου, στο Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ ε, έχει υποσχεθεί να είναι παρούσα. Η Κομισιόν, και η Κομισιόν ζήτησε αυτή τη μελέτη έτσι ώστε να ε, διαπιστώσουμε το πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ε, να υπολογίσουν το κόστος ε, των φαινομένων βίας κατά των γυναικών. Οπότε τι κάναμε. Εντοπίσαμε παρόμοιες μελέτες που έχουν γίνει όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν γίνει πολλές, αλλά σε χώρες παρόμοιες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαμε 10 τέτοιες μελέτες, βασισμένοι πάνω σε αυτές τις μελέτες αναλύσαμε ε, τα μοντέλα τους και την διαθεσιμότητα των στοιχείων. Έχουμε και εθνικές ε, και διεθνείς μελέτες. Είναι μια μελέτη η οποία, ε, την οποία θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο του χρόνου. έχουμε ένα ε, μοντέλο το οποίο βασίζεται στην ελάχιστη, στα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία ε, ε, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν οι διοικητικέ αρχές πάντοτε. Γιατί εξετάσαμε και το θέμα του τι στοιχεία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στις διοικητικέ αρχές. Ε, στις 8 Δεκεμβρίου λοιπόν θα ενημερώσουμε το Συμβούλιο για το θέμα αυτό των διοικητικών στοιχείων ε, των στοιχείων που διαθέτουν οι διοικητικέ αρχέ. Για παράδειγμα, εξετάσαμε τι κοινωνικέ υπηρεσίε, ε, τι υγειονομικέ υπηρεσίε, τη δικαιοσύνη και την αστυνομία. Όλε τι ε, δημόσιε αρχέ για να δούμε <clears throat> τι δεδομένα διακρατούνται, τι στατιστικές <clears throat> και είδαμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίε διαθέτουν πολλά στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών, οπότε αυτό είναι μια πρόκληση για μας του χρόνου να ξεκινήσουμε με τα κράτη-μέλη να ε, δουλεύουμε στο θέμα της εναρμόνισης των ορισμών. Γιατί ακόμα και οι ορισμοί διαφέρουν. Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται τα επεισόδια, ε, οι υποθέσει βία κατά των γυναικών είναι διαφορετικός, οπότε θα προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν το μακρόπνο, το μακρόπνο σχεδιασμό μας ε, του χρόνου. Ε, Θέλουμε ε, να κάνουμε μια χαρτογράφηση των μεθοδολογιών και των ενιών που σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων. Θα κάνουμε μια, ε, κάποιες συστάσεις ε, για καλές πρακτικές και τρίτον κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την αρμόνιση των δικτών ε, για τα θέματα της βίας κατά των γυναικών. τώρα έχουμε και την εκστρατεία της ε, Λευκής Κορδέλας. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου συμμετείχε, αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Ελπίζουμε ότι και άλλοι άντρες ε, ευρωβουλευτές θα μας υποστηρίξουν, όπως είπε ο κ. Ταραμπέλα σήμερα. Ε, οι άντρες ε, θα βοηθήσουν άλλους νεότερους άντρες και αγόρια ε, να ε, ανέβουν στο τρένο. Θα στείλουμε ξανά τις πληροφορίες λοιπόν στη γραμματεία και θα ζητήσουμε να ε, διανεμηθούν ευρέως. Θα θέλαμε και εσείς να συμμετάσχετε, είναι σημαντικό να σταλεί αυτό μήνυμα. Αυτές είναι οι συνεργασίες μας και τώρα πάμε στο mainstreaming την αρχή του 2015 θα ξεκινήσουμε, θα εγγενιάσουμε ένα ε, ηλεκτρονικό εργαλείο για το mainstreaming. Είπαμε σήμερα πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε παραδείγματα, να δίνουμε παραδείγματα ε, που δεν είναι παραδοσιακά ευαίσθηση ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων Έχουμε 9 τέτοια παραδείγματα, τα οποία θα ανεβάσουμε στο ίντερνετ, με την, ε, τον ορισμό, την περιγραφή για το τι, ποια είναι η σχέση ε, που εμπλέκεται η ισότητα των ε, φύλων. Έχουμε μεθόδους, καλές πρακτικές και κατάλογο οργανώσεων που ασχολούνται με την δημιουργία ικανοτήτων. Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα, τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικές διευθύνσεις κλπ. Τα ωφέλη της ε, ισότητας των φύλων. Θα ξεκινήσουμε μια μελέτη για να συλλέξουμε πληροφορίες ε, για τα οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της ισότητας. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να πείσουμε ακόμα και αυτούς που πιστεύουν ότι έχει ήδη επιτευχθεί η των φύλων. Να τους πείσουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να μαχόμαστε γι' αυτό. Ε, το κέντρο τεκμηρίωσης πριν από μερικά χρόνια αντιληφθήκαμε ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι όροι ε, ισότητας των φύλων δεν υπάρχουν καν στα λεξικά μας, τα ηλεκτρονικά μας λεξικά κλπ. Ε, ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το mainstreaming δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λέξη κλειδί, παρόλο που το χρησιμοποιούμε ε, στα ηλεκτρονικά εργαλεία. Οπότε μαζί με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και κάποιες ε, βιβλιοθήκες, ξεκινήσαμε και ελπίζουμε θα τελειώσουμε του χρόνου αυτή τη δουλειά, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα ορισμών, περιγραφών, ορολογίας. Πολλοί ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Γυναικών και πέρυσι και προηγουμένως είχαν πει ότι χρειάζονται ιδιαίτερες πληροφορίες για την ποιότητα των δεδομένων και μετά Έχουμε τη μεγάλη πηγή κοινή που είναι το κέντρο πηγών σε διάφορες γλώσσες, με διάφορες μελέτες, γιατί συνδεόμαστε με τα μεγαλύτερα κέντρα τεκμηρίωσης σε διάφορες χώρες. Φυσικά η διαδικασία κρατάει πολύ, έχουμε 10-12 χώρες μέλη, αλλά αυτό σημαίνει ότι με τη σύνθεση αυτή στον ιστό μπορούμε να με ένα κλικ να έχουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Για το Eurogender που είναι και αυτό ένα από τα καθήκοντά μας για την αξιολόγηση. Προσπαθούμε να δούμε οι συζητήσεις που κάνουμε, σε τι βοηθάνε, πού μας οδηγούν και θα δούμε και τι άλλα θέματα θα συμπεριλάβουμε. Το τελευταίο μου είναι ή διεθνείς δραστηριότητες. Να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη επιτυχία στη συνεργασία μας με τις χώρες προσένταξη. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Μία χώρα μέλος, η Σουηδία, ε, κάνει κάτι και τώρα εμείς με τις χώρες από την Ανατολική Ευρώπη θα έχουμε μία δίμερη συνάντηση στο κτίριό μας. Η Σουηδική κυβέρνηση λοιπόν θα αναλάβει τις χώρες αυτές για δύο μέρες και θα συζητήσουμε τους θεσμικούς μηχανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό η γνώση, το βάρος, ολόκληρος ο ρόλος των ε, φορέων που ασχολούνται με τη διάσκεψη του φύλου μπορούν να στηρίξουν αυτούς που δουλεύουν για τέτοια θέματα αλλού. Και διεθνείς οργανώσεις βέβαια, έχουμε εταιρικέ σχέσεις και συνεργασία μαζί τους. Το ΣΥΝΤΟ, η πλατφόρμα για δράση, η της Κομισιόν και αυτονών το έργο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με δύο λόγια είχα να σας πω. Αυτά σχεδιάζουμε να κάνουμε και αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπακ. Η παρουσίασή σας ήταν ιδιαίτερα εκτενής και έτσι μπορέσαμε και καταλάβαμε πόσο σημαντικό έργο κάνετε στο Ινστιτούτο σας. Ελπίζω ειλικρινά να φανεί χρήσιμο σαν εργαλείο εργασίας και στη δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Συζήτηση τώρα. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Λοιπόν, με τη σειρά. Πρώτον, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, η κυρία Λιγκέτσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά εσάς και το Ινστιτούτο, την Διευθύντρια, πρώτα απ' όλα την κυρία Λάμπακ, για την τόσο εκτενή παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου σας και τα μελλοντικά σας σχέδια. Το αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής δείχνει ότι πράγματι είναι αναγκαίο το Ινστιτούτο αυτό, γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία εμείς για τις 28 χώρες μέλη. Δεν έχουμε αρκετά τα οποία να μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πλήρως την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ακόμα και αν έχουμε τους δείκτες ισότητας των φύλων. Αν δούμε τα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη μέση του δρόμου σε σχέση με τον τελικό της στόχο, γιατί σύμφωνα με τους δείκτες είμαστε στο 54%. Συνεπώς, το Ινστιτούτο σας, όπως επίσης και άλλα ευρωπαϊκά όργανα, κάνουν πολλά και τους μένουν βέβαια ακόμα περισσότερα να κάνουν στο μέλλον. Εγώ προσωπικά προσβλέπω τη, στην εκδήλωση αυτή της 10ης Δεκεμβρίου. Ελπίζω να δω αρκετού συναδέρφους εκεί. Και ξέρετε ότι η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στην ενδοικογενειακή βία και στη βία κατά των γυναικών. Πιστεύω ότι μετά θα συζητήσουμε τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Θα συζητήσουμε επίσης την συνεργασία μας, η οποία πρέπει να επεκταθεί περισσότερο. Από τις πρόσφατες συζητήσεις και μάλιστα από αυτά που είπε και ο ίδιος ο Πάπας, ακούσαμε για τη βία, κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Τέλος, πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας και μαζί να καταπολεμήσουμε τη βία σε βάρος των γυναικών και να προσπαθήσουμε να υιοθετηθούν αποφάσεις. Θέλω επίσης να συγχαρώ το Ινστιτούτο σας για τη συνεργασία του με τα κέντρα τεκμηρίωσης. Πρόκειται για μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Εγώ θεωρώ ότι το βήμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί ευρέως και από και από ερευνητέ και τέλος τέλος από τους ίδιους τους πολιτικούς. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τις δραστηριότητές σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Για τα αποτελέσματά σας είναι πολύ σημαντικά σήμερα. Η κυρία Βάνα έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και σας κυρία Λάγκμπακ. Εγώ μίλησα και πριν για τη σημασία των στατιστικών στοιχείων και είναι πολύ σημαντική η δουλειά σας. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, αναφέρεται τον προϋπολογισμό και την ενσωμάτωση του φύλου. Έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, στατιστικά δεδομένα. Γιατί έθεσα ερώτημα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και μου είπανε δεν υπάρχουν δεδομένα, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε δεδομένα». Και είπα «Α, μα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας». Και μου είπανε το ποιο, οπότε το ερώτημά μου είναι ε, πώς θα διαδώσετε την ύπαρξή σας ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιο είδους μάρκετινγκ χρειάζεται γιατί καλή συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αλλά τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από όλους τους πολιτικούς ε, και να πάνε ειδικά σε αυτούς που δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για τα στατιστικά στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Παγκίνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λάμπακ για την παρουσίασή σας πολύ ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση έχω μόνο να κάνω. Από το Ινστιτούτο σας έχετε καμιά μελέτη για τις δημόσιες δαπάνες σε πολιτικές υπέρ των γυναικών σε οποιοδήποτε τομέα στις χώρες μέλη, ανά χώρα μέλος. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πρόεδρος, τελευταία η κυρία Νόης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ιδίως είναι άλλο να νιώθουμε ανισότητες και άλλο να το ξέρουμε ότι υπάρχουν, χρειάζονται άρα τα στατιστικά δεδομένα. Το ερώτημά μου είναι το εξής, μπορούμε να σας αναθέσουμε κάποια πράγματα. Εγώ ως βουλευτής, αν θέλω δεδομένα για κάτι μπορώ να σας δώσω, να σας αναθέσω κάτι. Muy bien. Creo que las... Καλώς. Οι ερωτήσεις σας ήταν πολύ συγκεκριμένες, νομίζω. Η κυρία Λάμπακ, λοιπόν, τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλές και συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις. Αν δεν μπορέσω να απαντήσω τώρα, θα σας απαντήσω σε μια εβδομάδα το πολύ, γιατί κάποιες ερωτήσεις όπως ε, το προϋπολογισμό για το φύλλο κτλ. Αυτό το οποίο προγραμματίζουμε είναι αυτό το οποίο θα ξεκινήσουμε μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε κάποιο θέμα σχετικό και επίσης αξιολόγηση αντικτύπου που είναι κάποιο είδους προϋπολογισμός, οπότε πράγματι για το θέμα της ενημέρωσης το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πράγματι είμαστε μόλις 4,5 ετών και πρέπει πράγματι να διαφημίσουμε την ύπαρξή μας. Και αυτό ακριβώς ε, συζητάμε τώρα, αλλά επίσης προγραμματίζουμε για το επόμενο έτος ε, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις πληροφορίες για τους διάφορους τομείς και να τα στείλουμε στις ε, διάφορες μονάδες πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς έχει σχέση το φύλλο με το περιβάλλον. Πώς σχετίζεται με την εκπαίδευση. Και τη σχέση με το δίκτυο. Βεβαίω θα έχουμε και το σχετικό link από κάτω, τον σύνδεσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες ε, πρωτοβουλίες. Έχουμε και την ε, έκθεσή μας για τους θεσμικούς ε, μηχανισμούς. Οπότε περιέχονται εκεί πέρα όλα αυτά, ενσωμάτωση του φύλου, ο προπολογισμό, αξιολόγηση αντικτύπου, κάποια άλλα παραδείγματα. Η Αυστρία είναι πάρα πολύ καλή στο θέμα αυτό του προϋπολογισμού για το φύλο. Και βέβαια ε, εξαρτάται και από τα αιτήματα των βασικών ε, ενδιαφερομένων μας. Οπότε ναι, πράγματι ε, μας ενδιαφέρει και απόψη σα, αλλά πρέπει να επικοινωνούμε τώρα για τη μελέτη πόσα ξοδεύονται για τις πολιτικές για τις γυναίκες στα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες γιατί, για να αναφερθώ και στο ερώτημά σας, ε, έχουμε αυτά τα βασικά καθήκοντα που είναι κομμάτι της ε, στρατηγικής της ε, Κομισιόν ε, και του κανονισμού για να έχουμε κάποια νούμερα, παραδείγματο χάρη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα στη συζήτηση, αλλά είχαμε τα εθνικά σχέδια δράση. Ε, είχαμε μια πάρα πολύ λεπτομερή εξέτασή του και εκεί πέρα βλέπετε το ότι υπάρχει όχι από πλευρά προπολογισμού, αλλά ποιε είναι οι προτεραιότητε των κρατών μελών, παραδείγματο χάρη για τα κορίτσια, για τα, την ηλεκτρονική παρενόχληση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δίνουν κάποια ιδέα, αλλά όχι ακριβώς ε, υπόμορφη προϋπολογισμού και μετά για συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό το οποίο κάνουμε συνήθως, μα γι' αυτό έχουμε αυτή την ε, βάση δεδομένων η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει μία απάντηση. Αν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα για την ισότητα θα υπάρχουν στην δικιά μας τη βάση δεδομένων. για να μας αναθέσετε μελέτη τώρα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τον προπολογισμό που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήθως οι δραστηριότητες ε, είναι προγραμματισμένες, ε, οπότε αυτό σημαίνει πως ε, για να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάτι εκτός αν είναι κάτι το τελείως αμεληταίο θα πρέπει να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι εκεί πέρα τα 19 κράτη-μέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα χρειαστεί λίγος χρόνος αλλά τα δεδομένα, πληροφορίες, όπως ανέφερε και η κυρία Μπλισκεβιτσιούτε, το κέντρο τεκμηρίωσης, όλα αυτά τα έχουμε, μπορούμε να τα δώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Σίγουρα θα μας ωφελήσει αυτό το, το έργο του Ινστιτούτου. Και όπως είπα και στην αρχή, ελπίζω θα πολλαπλασιάσουμε αυτές μας τις επαφές. Κλείνουμε για τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο στις 9. Έχουμε συνάντηση των συντονιστών και στις 10 θα ξεκινήσει η Επιτροπή.